Καλή σας ημέρα Αλφή, ας ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε όλοι παρόντες, αλλά η ημερήσια διάταξη μας είναι πολύ φορτωμένη. Ας ξεκινήσουμε το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού, του τρέχοντος ε, γενικού κανονισμού της ε, πολιτικής ε, στο πλαίσιο της εισαγωγής ενός καινούριου μέσου ε, μιας ε, καινούργιας ε, διευκόλυνση για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Το Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο συζητήσαμε τρεις φορές το ζήτημα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων οργάνων δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της ε, Task Force για την Ελλάδα. Ήταν εδώ ο πρόεδρος της Task Force ε, και μας μίλησε για τη σημασία αυτού του εργαλείου. Επίσης, ε, μας ενημέρωσαν σε τεχνικά briefing από πλευράς Κομισιόν και η οποία μας έκανε και γραπτές διευκρινήσεις, συναντηθήκαμε και με τους κοιόδους ηγητές, οπότε η συζήτηση αυτή έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο θέμα που να το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ ε, στην Επιτροπή μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το, το μέσο για χώρες όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερος. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση και η συζήτηση και θα καθοριστεί η ημερομηνία υποβολής τροπολογιών η 1η Μαρτίου. Η Επιτροπή μας θα ε, ψηφίσει τελικά το κείμενο στις 20 Μαρτίου, κάτι που θα μας επιτρέψει να στείλουμε το κείμενο στην Ολομέλεια του Απριλίου, έτσι ώστε η υπογραφή να λάβει χώρα τον Μάιο. Αυτό, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας, ελπίζω να μπορέσουμε να το τηρήσουμε. Στην πρώτη μας συνεδρίαση είχαμε συμφωνήσει, σα υπενθυμίζω, ε, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της ε, απλής ανάγνωσης, μονής ανάγνωσης. Διότι το θέμα επήγει. Το Συμβούλιο ξεκίνησε να συζητά το θέμα μόλις τον Ιανουάριο, συνεπώς ο χρόνος που έχουμε ε, για διαθεσμική συζήτηση είναι πολύ λίγος. παρόλα αυτά, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε συνένεση πολύ γρήγορα σχεδόν επί όλων των σημαντικών για μας θεμάτων. Οπότε η κατάσταση σήμερα είναι ως εξής. Το Συμβουλίο σε επίπεδο Κορεπέρ θα μπορούσε να υιοθετήσει το έγγραφο αυτό στις 14 Μαρτίου. Συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο έτσι ώστε να μην μπλοκάρει ο ένας τον άλλο χρονικά. Θα θυμάστε ίσως ότι η ιδέα πίσω από αυτή την τροποποίηση βασίζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Μεγάλα ε, project υποδομών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα υποδομών, είναι μπλοκαρισμένα εδώ και πολλούς μήνες εξαιτίας της ε, έλλειψης ιδιωτικής συγχρηματοδότησης. Αυτό το μέσο λοιπόν διαμερασμού του κινδύνου ε, διευκολύνει την πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα σε χρηματοδότηση. Πρόκειται ε, για project τα οποία, για τα οποία υφίστανται συγκεκριμένα οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την κρατική ενίσχυση. Συνεπώ, αν δεν εγκρίνουμε αυτό το μέσο, τότε αυτά τα project δεν θα μπορέσουν να ξεμπλοκαριστούν. Αυτό θα οδηγήσει βέβαια σε τεράστιες δημοσιονομικές συνέπειες για το ελληνικό κράτος γιατί θα χρειαστεί να πληρωθούν αποζημιώσεις στους ε, παραχωρησιοδόχους κλπ. Βέβαια, και οι τέσσερις χώρες που βρίσκονται σε ειδικό μακροοικονομικό καθεστώς ε, βοήθειας ε, μπορούν να υποφεληθούν του κειμένου αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία επίσης. Βέβαια, Προς το παρόν μόνο η Ελλάδα έχει εκφράσει τέτοιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε αν και οι άλλες τρεις ε, χώρες θα ζητήσουν να υποφελθούν. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις δεσμεύσεις ε, του 2012 του 2013 από την πολιτική συνοχής. Βέβαια, από του χρόνου και μετά η διαδικασία, θα αρχίσει να εφαρμόζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης. Ε, είχαμε διάφορα θέματα να αντιμετωπίσουμε, τεχνικά και νομικά. Καταρχήν, συνεργαστήκαμε πολύ με την νομική υπηρεσία, χρειάστηκε να τροποποιήσουμε πολύ την αρχική πρόταση της Κομισιόν, γιατί η αρχική πρόταση της Κομισιόν βασιζόταν στην υπόθεση ότι χρειαζόμαστε μία ε, ρήτρα διευκόλυνσης ε, και τις λεπτομέρειες θα τις ρυθμίζαμε σε ε, κατοπινές συμφωνίες. Όμως ε, χρειάστηκε να κάνουμε πολλές διευκρινήσεις στο κείμενο, ορίζουμε την διευκόλυνση διαμέσου του κινδύνου, τη συνδέουμε με το υπάρχον σύστημα των, του μέσου κατανομής του κινδύνου. Μιλάμε για πολλά στοιχεία της διαδικασίας. Δύο σημαντικά για το Κοινοβουλίο θέματα προέκυψαν. Να σας ενημερώσω για αυτά. Πρώτον, η γεωγραφική κάλυψη. Ποιες χώρες δηλαδή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε, αυτή την, σε αυτό το μέσο. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους σε όλες τις χώρες. Άλλοι επιθυμούσαν να περιοριστεί, όπως είχαν περιοριστεί και προηγούμενοι κανονισμοί, σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και που καλύπτονται από το σύστημα μακροοικονομικής ε, βοήθειας. Επίσης συζητήσαμε την ε, τεχνική δυνατότητα, ε, τις τεχνικές ικανότητες και δυναμικό της Κομισιόν να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι κάτι καινούριο, ενώ το Συμβούλιο που συζήτησε τα ίδια θέματα ε, εξέφρασε την ανάγκη, την επιθυμία να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πεδίο εφαρμογή, μόνο στην Ελλάδα ή δυνατόν. Οπότε τελικά καταλήξαμε στην ενδιάμεση λύση των προηγούμενων τροπολογιών. Έχουμε τις συγκεκριμένε χώρες οι οποίες καλύπτονται από συστήματα μικρονομική βοήθεια και μόνο αυτές οι χώρες θα μπορέσουν να ε, επωφεληθούν. Η Λετωνία και η Ουγγαρία δηλαδή δεν καλύπτονται από αυτό το μέσο. Συμφωνήσαμε λοιπόν <clears throat> για αυτό το θέμα. Για μένα αυτή η συμφωνία είναι απόλυτα λογική. Το δεύτερο θέμα ήταν ιδιαίτερα ακανθώδες και αφορά την επιλεξιμότητα συγκεκριμένων project. Και εδώ υπήρχαν δύο θέσεις. Η πρώτη θέση πρότεινε να περιορίσουμε το πεδίο των επιλέξιμων project στα project τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε η θέση ορισμένων συναδέλφων κυρίως του Κοινοβουλίου να καλύψουμε όλα τα project, όχι μόνο αυτά της πολιτικής συνοχής. Και πάλι είδαμε τα επιχείρηματα των δύο πλευρών. Το ένα επιχείρημα ήταν ότι η απόλυτη προτεραιότητα ήταν τα project της πολιτικής συνοχής γιατί εκεί είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς έχουν μια πιο πλατιά ε, ατζέντα project θα μπορούσε η χρηματοδότηση όλων αυτών να θέσει το περιθώριο τα project κοινωνικής συνοχής. Οπότε η θέση μας ήταν σαφές ότι θα πρέπει τα project να είναι project κοινωνικής, ε, συγγνώμη, πολιτικής συνοχής. Οπότε αυτά είναι απόλυτη προτεραιότητα. Βέβαια, δίνουμε τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν και σχέδια τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος ε, Αναφοράς, ο ΕΣΠΑ. Συνεπώς προτεραιότητα στα project πολιτικής συνοχής, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε και αυτά και να πάμε και σε project τα οποία ε, συνάδουν με τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή κάποιο οποιοδήποτε άλλο διεθνέ χρηματοπιστωτικό ε, φορέα η, χρηματοδότηση θα γίνει με βάση ε, κατά περίπτωση Ανάλυση και βέβαια στο πλαίσιο των κανόνων της χρηστής διαχείρισης. Νομίζω ότι ο συμβασμός που βρήκαμε ε, ανταποκρίνεται στην ανάγκη τα, να καλυφθούν κυρίως και καταρχήν τα project ε, της πολιτικής συνοχής. Όλα τα όργανα και οι ε, φορείς, ε, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δέχτηκαν τελικά το συμβασμό αυτό. Η, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δέχτηκαν το πρόγραμμα αυτό. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιότσιγητές τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένο με τις απαντήσεις που έλαβε από την αρχή της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Γιατί νομίζω ότι φτάσαμε σε μια κάποια συμφωνία που δεν ήταν προφανής από την αρχή. Η έκθεση είναι πολύ τεχνική, πολύ λεπτομερής, έχει πολλές τεχνικές ρήτρε, δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε αυτές, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παίζει το ρόλο της σε αυτό το χρηματοπιστωτικό όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε τον επόμενο 1,5 χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε και να σεβαστούμε την προθεσμία, όπως είπατε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει ε, σχέδια αυτή τη στιγμή προς εφαρμογή Επομένως, από πλευρά μα τουλάχιστον θα πρέπει να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να υιοθετηθεί αυτό το κείμενο τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Ε, κάνω έκκληση και στους συναδέλφου, λοιπόν να κάνουν μια προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, είμαι ικανοποιημένη με όλους τους ορισμούς. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή, ακριβώς για αυτό το θέμα δεν ήταν σαφές τι σήμαινε. Ε, δεν ξέραμε αν θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα το ξέρουμε. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που το πετύχαμε. Μία ερώτηση μόνο έχω προς την Επιτροπή. Μια σύντομη ερώτηση για την τροπολογία 9 εκεί που μιλάμε για τους ε, εθνικούς φορείς ε, δημόσιας παρέμβασης. Όχι τους άλλους φορείς, αλλά αυτούς ειδικά που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Υπάρχει τέτοια βούληση από τέτοιους φορείς ε, να συμμετάσχουν. Υπάρχει κάποια ένδειξη. Σε, υπάρχει τέτοια διάθεση συνεργασίας σε τέτοιου είδους σχέδια, σε τέτοιου είδους project την επόμενη χρονιά. Η μόνη διευκρίνηση που θέλω να ζητήσω είναι αυτή. Κατά τα λοιπά δεν έχω άλλε ερωτήσει. Έχουμε συναντηθεί τόσε φορέ ούτω ή άλλω με του ενδιαφερόμενου. Όλοι οι σκιώδει, τα μέλη τη τράπεζα, οι κομισιόν ε, και θέσαμε ερωτήσει και όλε οι ερωτήσει που είχα και απορίε απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών. Η Ραμόνα Μανέσκου δεν είναι εδώ. Εκ μέρου των φιλελεύθερων, παρακαλώ είχαμε μεικτή, δηλαδή ο ένας είχαμε και δύο αρμοδιότητα και, και οι δύο είχαμε, λοιπόν, συμμετείχαμε. Μία ερώτηση προς την εισηγήτρια θέλω να κάνω. Οι χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να ζητήσουν την ενεργοποίηση αυτού του μέσου, είναι σαφές ποιες θα είναι. Αρχικά είχαμε πει ότι ήταν οι χώρες που είχαν πρόβλημα να βρουν κονδύλια. Αλλά τα προβλήματα μπορεί να είναι ποικίλα. Μπορεί να σημαίνει ότι οι τράπεζε δεν δίνουν. Μπορεί να σημαίνει ότι η διαχείριση σε αυτέ τι χώρε δεν είναι καλή. Ή ότι ο Υπουργό Οικονομικών στη χώρα αυτή είναι αδρανής, δεν κάνει τίποτα. Είναι μόνο η οτι ο υπουργο οικονομικων στη χωρα αυτη ειναι δρανης Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση προ την εισηγήτρια είναι εξή. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν διευθυντή Τράπεζα εγώ. Και τότε θεωρούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, δεν θα συγχρηματοδοτήσει απλώς, αλλά θα μπει και εγγυητής. Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει εγγυήσεις σε εμπορικές τράπεζες, οι οποίες αυτές δίνουν τα χρήματα. Και υποτίθεται ότι αυτή η εμπορική τράπεζα στη χώρα θα πρέπει να κάνει όλη την πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι η Τράπεζα Επενδύσεων θα κάνει παράλληλη και αυτή πραγματογνωμοσύνη ή θα ζητήσει κάποιες εγγύησεις, εμπράγματες εγγύησεις, σε κάτι, στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Γιατί αν πάει κάτι στραβά, τότε θα πρέπει να αναλάβει ένα τεράστιο κόστος η θα ζητησει καποιες εγγυησεις εμπραγματε εγγυησεις σε στην περιπτωση που κατι παει στραβα αυτή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Επενδύσεων δηλαδή. Σας ευχαριστώ για τις ε, δηλώσεις σας. Είχα δώσει γραπτά στη συνεργατή μου, γιατί δεν μπορούσα να είμαι χθε εδώ παρούσα. Είναι πάντως αφή η θέση μας. Το μέσο αυτό το υποστηρίζουμε, αλλά έχουμε επιφυλάξεις ε, λόγω της διευκόλυνσης χρηματοδότησης των σχεδίων να χρηματοδοθούν και παράλογα σχέδια και γι' αυτό θα θέλαμε, τουλάχιστον για εκείνα τα σχέδια τα οποία είναι εκτός του κανονισμού να προβλεφθεί ο απαραίτητος έλεγχος για να εξεταστεί κατά πόσον είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά το όφελο στην δημοκρατική συμμετοχή των κατοίκων κλπ. Θα υποβάλουμε η ίδια τροπολογία. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek. já se domnívám, že je, je možné pomoci státům. Κατά τη γνώμη μου, ε, χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να βοηθηθούν με συγκεκριμένες ε, στοχευμένες επενδύσεις. Ξέρουμε ότι οι χώρες αυτές έχουν το πρόβλημα να βρουν ιδιωτική χρηματοδότηση. Βέβαια, υπάρχει κάποιος τρόπος βοήθειας δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσει εδώ να συμμετάσχει. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα επενδεθούν οι πόροι που θα δοθούν, αλλά θα πρέπει τα σχέδια που μεταδοθούν να είναι πολύ στοχευμένα και να έχουν σαν σημείο προσανατολισμού την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της απασχόλησης και την δυνατότητα της χώρας να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η επιλογή των σχεδιών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Lambert ε, van Ήμουν στην Επιτροπή Ήτρε. Ίσως κάτι να χάσα. Αλλά μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες στο Συμβούλιο ε, ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Για την νέα περίοδο λοιπόν 2014-2020 προβλέψαμε μια σειρά από μέσα, από εργαλεία όπως αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας. Αν θυμάστε τις συζητήσεις που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας, Είχε τεθεί το ερώτημα αν ε, θα ήμασταν έτοιμοι εγκαίρως να προσαρμόσουμε τον ισχύοντα κανονισμό. Πριν την έναρξη δηλαδή της νέας περίοδου. Γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο. όταν βλέπω τις ικανότητες απορρόφησης στις χώρες που έχουν πληγεί πιο έντονα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, έχω την αίσθηση ότι αυτό το μέσο παραμένει αναγκαίο, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον μοχλό βοήθειας. Χθες διάβασα σε μια εφημερίδα ότι ο Μπαρόζο μίλησε για την ενίσχυση των ε, μέσων ε, υπέρ της Ελλάδας. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει συγχρηματοδότηση. Και ίσως με τέτοιο τύπο εργαλεία έχουμε λιγότερο περιθώριο. Αλλά ας προσπαθήσουμε να είμαστε θετικοί. Ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το λέω αυτό ε, εν ονόματι της ομάδας μου, η οποία έχει αντίρρηση στην αρχή. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Είδα εξάλλου και μία, ένα κείμενο μάλλον της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Είναι ένα έγγραφο της 27ης Φεβρουαρίου. Τι Φεβρουάριο. Είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή, πολύ φρέσκο. Είναι ίδια φιλοσοφία και εκεί, αυτή που διέπει το έγγραφο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι κάθε ευρώ να ξοδεύεται με αυστηρές ε, προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, να υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το αποτέλεσμα να είναι αυτό. Θα πρέπει κάθε ευρώ να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές τις χώρες ε, με οικονομικές δυσκολίες. Όντως, η καιρή είναι χαλεπή. Θα πρέπει να βρεθεί μια νέα προσέγγιση από πλευράς κομισιών. Εγώ είμαι για το εξής. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτό το μέσο και μην ξεχνάτε και τη συζήτηση που κάνουμε με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί από πλευρά τους. Θα συνεχιστεί η συζήτηση, το λέω, και στρέφουμε προς τις άλλες ομάδες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι η Επιτροπή Ρέτζι να είναι έτοιμη να παραθέσει επιχειρήματα. Γιατί αλλιώς μπορεί η ομάδα μου ή άλλες ομάδες να προτάξουν πραγματικές αντιρρήσεις. Όντως προχωρούμε, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που ακριβώς θέλουμε. Ευχαριστώ. Κέλλη. Τζιν Κέλλη. Χαίρομαι για τις εξελίξεις γιατί τα κράτη-μέλη και ο τύπος μιλάνε πολύ έντονα για τα προβλήματα ε, λιτότητας. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόληση και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Μία ή δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Από ό,τι ξέρω, είναι τμήμα από αυτό των 82 δισεκατομμυρίων που είχαν ε, ανακοινωθεί πέρυσι ε, με σκοπό να δημιουργηθούν περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Η κυβέρνηση πρέπει να τα ζητήσει. Και γιατί project μιλάμε εδώ πέρα. Ενέργεια ας πούμε. Για μια χώρα σαν την Ιρλανδία ας πούμε. Που είναι υποτίθεται πλούσια σε, σε όρους ΑΕΠ. είναι κάτι παραπάνω από αυτό που εμείς έχουμε φύγει ουσιαστικά από το, το Ταμείο Συνοχής ε, και επομένω ε, επομένως αυτά τα λεφτά θα έρθουν να τα αντικαταστήσουν τα λεφτά της Συνοχής. Και επίσης ε, τα λεφτά αυτά μιλάμε ε, ότι θα δοθούν και μετά το 13, το 14 και το 15 δηλαδή. Ο επόμενος ομιλητής. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ χρήσιμη και επίγουσα αυτή η συζήτηση. Ε, για πολλές χώρες μεταξύ αυτών και την Ελλάδα πρέπει κατεπηγόντως να υφετηθούν μέτρα για να μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης, αλλιώς θα συζητιέται το θέμα μέχρι την Αγίων ποτέ. Υπάρχουν τρει λόγια γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό απορρόφηση σε ορισμένε χώρε. Καταρχήν, έλλειψη γνώσεων από του δικαιούχου. Και εκεί χρειάζονται μέσα ενημέρωση βέβαια. Κατόπιν, η έλλειψη των πόρων συγχρηματοδότηση, αυτό το συζητήσαμε διαμακρών. Είναι δύσκολο, όσο πάει και πιο δύσκολο μάλιστα να έχει κανένα πρόταση σε χρήματα για εξωτερική χρηματοδότηση. Επίσης το θέμα της γραφειοκρατίας που δεν έχει ζητηθεί τόσο πολύ και θα ήθελα να ξέρω τι πρόκειται να γίνει σχετικά με το θέμα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όσον αφορά τα παλαιά ποσά αυτά. Σε ορισμένε ε, περιπτώσεις έχουμε διαφάνεια, άλλες όχι. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Θα καταφέρουμε εμείς ε, να απλουστεύσουμε τους κανονισμούς ούτως ώστε να μπορούν τα χρήματα αυτά να φτάνουν στους δικαιούχους και να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ε, πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Thank you very much. I don't have any other speaker. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Παρακαλώ, μπορείτε να μας απαντήσετε τεχνικά θέματα και μετά εγώ θα παρέμβω για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Πριν απαντήσω στις τεχνικές ερωτήσεις, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας με την σημαντική πρόοδο που σημειώσαμε στα πλαίσια του Συμβουλίου τελευταίως. Χαίρομαι και για τις προσπάθειες που καταβάλλεται από πλευράς Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Από πλευράς Κομισιόν υποστηρίζουμε τον τρέχοντα συμβιβασμό Πιστεύουμε ότι είναι ισορροπημένος. Ισορροπημένη είναι η πρόταση. Λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που είχαμε εντοπίσει στη διάρκεια της συζήτησης. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία του μέσου αυτού και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ιδίως σε ό,τι αφορά το εύρος των project που υποστηρίζει αυτό το μέσο. Πρόεδρε, να προσθέσω και κάτι ακόμα που προέκυψε στη τελευταία συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου, που είναι η δημοσιονομική επίπτωση. Από πλευράς Κομισιόν δεχτήκαμε ότι θα υπάρξει κοινή δήλωση με το Συμβούλιο για θέματα περιορισμού της δημοσιονομικής επίπτωσης του μέσου αυτού. Στον κανονισμό έχουμε κάποια, κάποιες παραμέτρους ελέγχου που πιστεύουμε ότι εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το 10% που είναι ε, διαθέσιμο για ένα κρατός μέλος. Ε, για την ετήσια προετοιμασία του προϋπολογισμού όμως θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα, αναταράξεις κτλ. Και τις ερωτήσεις η κυρία Κλέμπερ ρώτησε αν υπάρχουν και άλλοι διεθνείς φορείς ε, που ενδιαφέρονται ε, να επιμεριστούν αυτό το κίνδυνο στα πλαίσια της Ελλάδας. Έγιναν συζητήσεις σιγά, οι οποίες συνεχίζονται ούτως ώστε να φέρουμε και άλλες διεθνείς ε, τράπεζες, όπως την KFW από τη Γερμανία. Αλλά όπως έχει συζήτηση αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε όμιλος ή consortium που μπορεί να δημιουργηθεί ως επενδυτής μπορεί να είναι έτοιμος να συμμετάσχει στα πλαίσια του μέσου όπως έχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι Κυρίω θα είναι δουλειά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εφαρμόσει την πρόταση αυτή α, του επιμερισμού του κινδύνου για την Ελλάδα καταρχήν. Ο επόμενος ομιλητής έκανε μία ερώτηση ε, για τις εγγύησει. Μην ξεχνάτε το εξής, ότι η συνεισφορά από την εθνική συνεισφορά της εν λόγω χώρας θα βγει από τα επιχειρησιακά προγράμματα και θα πάει σε αυτό το μέσο. Και οι εγγυήσει θα είναι ένα κεφάλαιο για τις δράσεις που θα δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με άλλους φορείς, τράπεζες, ε, αναδόχους ή οποιονδήποτε άλλο ε, από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια ως ένα κεφάλαιο, ας πούμε, ως μια εγγύηση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά στο οποιοδήποτε project, στο οποιοδήποτε σχέδιο. Προσπαθούμε να ελέγξουμε τον κίνδυνο με μεγάλη αυστηρότητα. Συμφωνήθηκε ότι όλα τα project θα ελεγχθούν πολύ σωστά, ούτω ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος θα ελεγχθούν λοιπόν με κάθε επιμέλεια, με κάθε αυστηρότητα. Η κυρία Σρέντερ έκανε μια ερώτηση για project που εκφεύγουν του NSRF, που δεν έχουν δηλαδή άμεση συνδρομή από την περιφερειακή πολιτική. Είναι σε μια δεύτερη ας πούμε κατηγορία. που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής, που προωθεί τους στόχους δηλαδή της πολιτικής συνοχής. Αλλά δεν έχουν άμεση οικονομική συνάφεια. Πιστεύουμε ότι επειδή αποφασίζουμε εξατομικευμένα για κάθε σχέδιο και επειδή έχουμε και κάποιες τεχνικές ε, προϋποθέσεις, μπορούμε να ελέγξουμε και την ποιότητα που θεωρούμε απαραίτητη για αυτά τα σχέδια τα οποία θα λάβουν ε, βοήθεια, οικονομική βοήθεια μέσα από αυτό το εργαλείο που δημιουργούμε. Ο κύριος Κέλλη μίλησε για την ε, ανακατανομή των πόρων και αν έχει καμία σχέση με το, αυτή η κατανομή, με αυτό το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Όχι. Γιατί αυτά τα 82 δις που ανέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν, αφορούν ποσά που δεν έχουν ακόμη δοθεί σε συγκεκριμένα project στην πολιτική συνοχής. Φυσικό είναι αυτό. Δεν έχουν επιλεγεί ακόμα όλα τα project. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι ένα μέτρο κρίσης, διαχείρισης της κρίσης. Άλλο είναι η ανακατανομή ή ο επαναπρογραμματισμός κονδυλίων. Στα πλαίσια της επιλογής των project. Τώρα, τι είδους project ναι, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς αυτά είναι project τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν από αυτό το μέσο. διότι ευθυγραμμίζονται πλήρω με τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Τέλος. Πόσο διαρκεί η χρηματοδότηση. Όταν δημιουργηθεί αυτό το ταμείο, θα ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο. Δηλαδή θα ξεπεράσουμε και το 2015, σίγουρα. όπως και στην περίπτωση άλλων τέτοιων μέσων, στο τέλος θα πρέπει να αποδείξουμε ότι όλα τα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί ή παύλα επενδυθεί για project. Καθόλου δεν θα πρέπει να δοθούν χρήματα για project, για σχέδια μη επιλέξιμα. Να προσθέσω και εγώ μερικά λόγια. Θα θυμάστε στις δύο προηγούμενες τροπολογίες ε, Αυτές αποτελούσαν ε, αποτέλεσμα της απόφασης Συμβουλίου ότι οι έξι χώρες που καλύπτονται από τα συστήματα μακροοικονομικής ενίσχυσης ε, θα έπρεπε να δοθούν ε, τέτοιου είδους ε, εργαλεία για να βελτιωθεί η ανάπτυξη. Μέσα σε αυτές τις χώρες βρισκόμαστε, αλλά όχι όλες πια, γιατί η Ουγγαρία, παράδειγμα, και η Λετωνία έχουν πλέον εξαιρεθεί. Η Ουγγαρία και η Λετωνία δεν ενδιαφέρεται, οπότε έχουμε τέσσερις μόνο. Μετά, η Κομισιόν... Ε, το 2006 ξεκίνησε το Τζέρμι και το Τζέσικα με την, ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τότε μπήκε και η KFW. Ήταν η μόνη τράπεζα η οποία ενδιαφέρεται, είναι η μόνη που ενδιαφέρεται ακόμα. Δεν έχουμε καμιά άλλη που να ενδιαφέρεται. Τώρα σε ό,τι αφορά την ανάγκη αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί και για την πρόθεση απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, ε, έτσι κι αλλιώς ε, θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού σημαντικά τεράστια εθνικά project υποδομών, συνεπώς σίγουρα θα ενεργοποιηθεί η οικονομία και θα δημιουργηθεί θέση εργασίας. Τώρα, αν στην Ελλάδα θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση, όχι, υπό την έννοια ότι θα έρθουν περισσότερα χρήματα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όμως είναι ε, περισσότερα χρήματα διότι χρειάζεται η ε, μόχλευση και με τον τρόπο αυτό, μέσω αυτού του σχήματος έλκουμε και περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Συνεπώς αυξάνονται τα συνολικά κεφάλαια. Τώρα, μιλούμε για δύο δόσεις δεσμεύσεων. Τα φετινά, τη φετινή δόση και την επόμενη του χρόνου. Οπότε στο μέσο του επόμενου χρόνου περίπου θα πάψουν να είναι διαθέσιμα ως δεσμεύσεις αυτά τα χρήματα. Μέχρι τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μετά, Πετ Λούχαν, ε, δεν έχουν σχέση με αυτό ακριβώς το project, αλλά αυτό λέγαμε όταν συζητούσαμε το νομικό πλαίσιο για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Το θέμα είναι η απλοποίηση. Σίγουρα θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια... Α, σαν. Εφαρμόζεται μόνο στα κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχει πακέτο διάσωσης. Και αν αυτές οι χώρες στραφούν σε αγορές, το μέσο αυτό θα πάψει να χρησιμοποιεί. Επαναλαμβάνω, ε, αυτό καλύπτει μόνο τις χώρες που βρίσκονται σε πακέτο διάσωσης και αν κάποια αυτές οι χώρες επιστρέψει στην αγορά, στις αγορές. Τι θα είναι, θα πάψει να τις χρηματοδοτεί αυτό το μέσο. Δυστυχώς η, ομιλή, πρόεδρος μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Ε, αυτό το μέσον Ε, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μια χώρα μπορεί να αρχίσει να το χρησιμοποιεί όσο βρίσκεται σε καθεστώς μακροοικονομικής ενίσχυσης. Ε, πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν να το χρησιμοποιεί ε, όσο βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Από εκεί και πέρα μπορεί να βγει οποιαδήποτε στιγμή. Ίσως θα ήταν συνετό την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις τροπολογίες. Να ξαναφιερώσουμε λίγο χρόνο στην Task Force που εργάζεται για την Ελλάδα. Για να δούμε πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο. Γιατί όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ωραία, το κάθε μέσο έχει τις δυνατότητές του. Αλλά χτες άκουσα, για παράδειγμα, ότι ο Μπαρόζο ε, είπε, δήλωσε πως ε, είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει καινούργια μέσα για την Ελλάδα κλπ. Το θέμα είναι όμως ε, πού, πού, θα χρησιμοποιηθεί, σε τι project θα χρησιμοποιηθεί. Είναι δυνατόν να ξανακούσουμε την ομάδα για την Ελλάδα. Ε, μα, ε, πρόεδρος, ε, μα το κάναμε αυτό ήδη. Τους προσκαλέσαμε. Είδαμε, είχαμε εδώ το πρόεδρο της Task Force για την Ελλάδα, τον κύριο Ράχενμπαχ. Και θυμάστε, ότι συζητήσαμε το θέμα του ποια project θα χρηματοδοτηθούν. Μήπως θα μπορούσε να μας απαντήσει γραπτός. Ε, μα είπε, εντάξει, ωραία τα λόγια του, έπε απτερόεντα όμως. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πιστεί ακόμα. πώ θα μπορούσαμε να τους πείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα-δύο άτομα στην ομάδα μα. Ωραία, θα το κάνουμε. Και θα ζητήσουμε και από την Κομισιόν να μα υποβάλει γραπτός ε, τι είδου project θα καλυφθούν. Ξέρουμε ότι πρόκειται για αυτοκινητόδρομου, για ε, κομματερές, χιτά κλπ. Ε, αν δεν υπάρχουν σχόλια, προθεσμία για τροπολογία 3 το απόγευμα 1η Μαρτίου. Και να περάσουμε στις ψηφοφορίες παρακαλώ. can we... Αγαπητοί συνάδελφοι, για να ελέγξουμε, can we check... για να ελέγξουμε τα μηχανήματα, ε, τοποθέστε παρακαλώ τις κάρτες τα μηχανήματα να δούμε αν όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Ho dimenticato la carta di voto. Ξέχασα την κάρτα μου. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay we are waiting uh, for whoever is not yet ready. Λοιπόν, περιμένουμε. Θα αρχίσουμε στις 10 ακριβώς να ετοιμαστούν όλοι. Okay, αυτό Um, I, can we, can, is EPP ready to... In έτοιμο το ΕΛΚ. Is... Uh, can we start voting? So we check the... Μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Να ελέγξουμε τα μηχανήματα πρώτα. Έχουμε πολλούς που θα πρέπει να ψηφίσουν, αλλά δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Πιέστε τα κουμπιά εκεί. Εκείνοι που είναι νέοι και δεν έχουν ξαναψηφίσει, ίσως μπορούν να βοηθηθούν από τους γείτονες. So those colleagues who forgot the card have to signal. Όποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του πρέπει να πει στη γραμματεία πώ θα ψηφίζει εξάστοτε. Αρχίζουμε με την έκθεση τη Κατρίν Βέρντερ για την ασφάλεια ζωή το φυσικό μα κεφάλαιο και την βιοεπικοινότητα. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τα γλωσσικά, τις γλωσσικές τροπολογίες. 19 υπέρ, κατά, Αποχές. Να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρασε ψηφοφορίες. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα απορρίφθηκε. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άθλη ψηφοφορία. Uh, we close the vote. Πέρασε ψηφοφορίες. Ψήφισαν όλοι. 38 υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην συγγετρία, στην Κατρίν. Και περνάμε τώρα στο σημείο 12 είναι η έκθεση Thomas Deutsch για την απαλλαγή 2010. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3.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 αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας 38 υπέρ και 2 κατά συγχαρητήρια ενεκρίθη λοιπόν και περνάμε στην, ε, στο έκτο πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον, σήμερα 13, η συνάδελφο Ζωρίσα Διορίσα Ντάντσιρα στην συντάκτρια. Τροπολογία ε, συμβαστική υπέρ. Ένα. Α, όχι. Υπάρχει μια σύγχυση για να δούμε. Συμβαστική τροπολογία 1. Παρακαλώ. Είσαστε υπέρ. Ωραία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. 38 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Uh, so... Now we go on with, uh...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 για τους ε, κοινό κανονισμό και ένα μαντέρι ήταν τελευταία που υπέβαλε θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση σημείο 9 και θα δώσουμε το λόγο στην Κοντάντσα Κρέλ αλλά μην ξεχάσετε ότι έχουμε και μία σειρά άλλων κανονισμών σήμερα ζητώ συγγνώμη δεν μπόρεσα να προετοιμαστώ, δεν είμαι καθόλου καλά, δεν έχω τίποτα να σας πω. Σε ένα τέταρτο πρέπει να είμαι στον, στο γιατρό. Δείξτε κατανόηση μια φορά. Ο Λάμπερτ νομίζω θα με αντικαταστήσει πολύ καλά. Okay, so I understand that... Ναι, κατάλαβα. Ο Λαμπέρ λοιπόν θα είναι επικεφαλής της συζήτηση. Ωραία. Ωραία. Κάρι Μαντελ είχε υποβάλει μια ερώτηση αλλά δεν πήρε απάντηση από το Λαμπέρ νομίζω στις ανησυχίες σας για αστικά θέματα δεν κάνω λάθος Συζητήσαμε τρία θέματα χθε όσον αφορά το γενικό κανονισμό που ήταν το απόθεμα για την για τις επιδόσεις και διάφορα άλλα θέματα ε, είχαμε διακόψει και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε σήμερα. Αν κανένας όμως δεν θέλει να συνεχίσει σήμερα, δεν θα επιμείνω. Για τρία σημεία μόνο του Γενικού γνωσμού τα αστικά θέματα ε, μας ζήτησε ο Γιάννα που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, να τα συζητήσουμε την επόμενα. Λοιπόν, υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να θέσουν κάποιες ερωτήσεις για τα θέματα που συζητάγαμε χθε. Παρακαλώ, κ. Uh, Ζητώ συγγνώμη που ήμουν απόν στην απογευματινή συνεδρίαση χτες. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό επιδόσεων. Πρώτον, κατά την άποψή μου, θα το γράψω μάλλον, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό, Δεύτερον, λείπουν τα κριτήρια, κάτι που δημιουργεί τις συνθήκες για υποκειμενικές δράσεις, κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Και τρίτον, γιατί να τιμωρούνται με αυτόν τον τρόπο οι διάφοροι φορείς. Νομίζω ότι και η Επιτροπή των Περιφερειών είπε πως το απόθεμα αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί καλύτερα για να γίνει αποδεκτό. Για το ανώτατο όριο, το cupping, την οροφή. Με την οροφή είναι σαφές ότι μειώνουμε δραστικά τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής. Με την ε, δραματική μάλιστα μείωση του ΑΕΠ των κρατών μελών, η οροφή το μόνο που θα κάνει θα είναι να μειώσει τις, ε, ε, κονδύλια που ρέουν προς τα κράτη-μέλη της πολιτικής συνοχής. Με αυτόν τον τρόπο η πολιτική συνοχή θα γίνει κενή, κενός λόγος, κενή κουβέντα. Σε ό,τι αφορά το Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, ε, έχω κάποια προβλήματα με τις προτάσεις Κομισιόν, αλλά να σας πω το εξής ε, εδώ πέρα. Υπάρχει μια δραματική σαφής και δραματική ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού της σχέσης ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Κομισιόν και της κεντρικής κυβέρνησης στην επιλογή των project. Η βασική μου ανησυχία είναι αυτό το βιβλίο, όχι η δική μου προσωπική άποψη. Αυτό το βιβλίο ε, το, το, μας το παρουσίασε η DG Move στην Ανβέρσα Πρόκειται για προσχέδιο βέβαια, <laughs> αλλά βλέποντας τις προτάσεις υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν κανένα λόγο να είναι χαρούμενα με αυτές τις προτάσεις. Λοιπόν, καλύτερος ορισμός και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις αν θέλουμε να γίνει δεκτό αυτό το όργανο. Αυτές προτάσεις. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Yes. Για αυτά τα τρία θέματα, Σρέτερ, Τέλη κλπ για το Capping, το Connecting Europe και τα αποθέματα. Ναι, Πρόεδρε. Ένα σχόλιο πολύ σύντομα για τα τρία αυτά σημεία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο performance reserve, στο απόθεμα της απόδοσης. Εμείς θέλαμε να έχουμε μία ενίσχυση που προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί ούτως ώστε να πετύχουμε αυτή τη συμπληρωματική ενίσχυση, γιατί μάλλον συμβολικό χαρακτήρα έχει. Το κεντρικό πρόβλημα είναι πώς, ποια μορφή θα έχει ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και ποιοι θα είναι οι δείκτες που θα πρέπει να αναπτύξουμε. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πρόβλημα. Δεν είναι σαφές και γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές επικρίσεις. Και γι' αυτό αυτό το θέμα του αποθέματος απόδοσης θα πρέπει να το αναβάλουμε και να το εξετάσουμε με το θέμα της διατύπωσης των λειτουργικών σχεδίων. Αυτό που δεν είναι σαφές και στη διατύπωση γιατί κάθε υποκανονισμό έχει διαφορετική διατύπωση, είναι αυτά τα επίπεδα, δηλαδή η σχέση μεταξύ των αξώνων προτεραιότητας, των επενδυτικών προτεραιοτήτων και πώς θα μπορούμε αυτά τα διάφορα επίπεδα να δούμε πώς σχετίζονται με τους δείκτες που δεν είναι στο γενικό κανονισμό, είναι στους ειδικούς κανονισμούς. Αν τα έχουμε ε, διευκρινίσει όλα αυτά τα σημεία, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα του ε, performance reserve. Γι' αυτό κύριε Λαμπέρ, νομίζω θα ήταν καλύτερα να διευκρινίσουμε αυτή τη δομή με την Κομισιόν. Γιατί την έχει πολύ περιπλέξει αυτή τη δομή η Κομισιόν. Και αυτό που λένε ορισμένοι τώρα ότι παρά είμαστε ε, γραφειοκράτες ε, είναι σωστό. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε το θέμα με την Κομισιόν. Να δούμε ποια είναι αυτά τα επίπεδα και τι θα γίνει με τους διάφορους δείκτες. Δηλαδή αυτό το απόθεμα απόδοσης που θα ξεκινήσει ανάλογα με το αποτέλεσμα με τους δείκτες δηλαδή αποτελέσματος ή με κάποιο άλλο τρόπο. Μόνο εάν αυτό το θέμα διευκρινιστεί θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα της performance reserve γιατί θα είναι ξεκάθαρο από πού ξεκινά και από πού όχι. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το συζητήσουμε αργότερα όταν έχουμε ε, διευκρινίσει πώς προβλέπει η Κομισιόν τον προγραμματισμό. Thank you very much. I would just like to inform... Ευχαριστώ να ενημερώσω τους αδέλφους που ήταν απόντες ε, χτες το πρωί όταν έγινε η παρουσίαση της κυρίας Πελεγκρέ από το κέντρο ε, βιομηχανικών σπουδών του Μιλάνου για την ε, πολιτική που είναι προσαρμοσμένη στις επιδόσεις υπάρχει μια μελέτη η οποία αναφέρει πάρα πολλά πράγματα ε, και μπορείτε να τη διαβάσετε. Κάριμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω στο Urban. Αλλά να σας πω τι εγώ δεν καταλαβαίνω. Καταρχήν, η διακυβέρνηση. Η Κομισιόν λέει ότι έχουμε φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Πώς φτάσανε στα 10 δισεκατομμύρια, ποια ήταν τα κριτήρια, πώς θα καθοριστούν οι άξονες προτεραιότητας. Έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν μέσω μιας ε, διακυβέρνησης ε, από κάτω προς τα πάνω λέει αμφισβητεί την, το δικό μας σύστημα, αυτό το σύστημα που έχουμε προτείνει εμείς και θα ήθελα να μου δώσει τη γνώμη του και ο κ. Φανλής γι' αυτό. Γιουνούς. Καταρχήν μια γενική παρατήρηση. Χαίρομαι που βλέπω ότι και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο διαμορφώνεται μια κατά συνένεση για τα βασικά. Αυτό θα μας ενισχύσει, θα ενισχύσει τη θέση μας στις συζητήσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Μία παρατήρηση για το αποθεματικό απόδοσης. Πρόκειται για ένα ε, βαθιά άδικο μέσο που μας απομακρύνει από την αρχή της ε, ε αλληλεγγύης. Νομίζω ότι ο κ. Φανίστελ Ρόιτ το υπογράμμισε χτες. Διαφωνούμε με αυτή την πρόταση διότι ε, εξομοίωνουμε αυτή την πολιτική με την πολιτική του καρότου και του μπαστούνιου. Η Κομισιόν δεν καταφέρνει να μετρήσει την απόδοση έτσι κι αλλιώς, ούτε και να καθορίσει τις πραγματικές προτεραιότητες. Και δεν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό στη θέση των περιφερειών. Οι περιφέρειες μόνο μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε ε, το απόθεμα αυτό ε, γίνεται τελικά απόθεμα καλής διαχείρισης και όχι απόθεμα απόδοσης. Οπότε <laughs> και το ερώτημα που είναι τι θα γίνει με τα αποθέματα τα οποία δεν θα έχουν ε, εκταμιευθεί. Θα εκταμιευθούν σε άλλα κράτη. Δεν μου φαίνεται πολύ δίκιο Ούτε και σύμφωνο με την αρχή της συνοχής. Η απόδοση θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ των υστέρων και θα πρέπει να επηρεάσει τις στρατηγικές. Συγγνώμη. Ε, η απόδοση θα πρέπει να μετρηθεί εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Ε, η απόδοση με τη μέτρησή της θα πρέπει να επηρεάσει το σχεδιασμό των πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα χθε. Ήμουν σε μια άλλη επιτροπή όμω. Συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε γενικά σήμερα για, ε, το αποθεματικό απόδοση που έχει εισαχθεί. Πρέπει να ξαναδούμε την ε, δική μας θέση. Όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, όταν θα γνωρίσουμε περισσότερα τα κριτήρια που σκοπεύει να υιοθετήσει η Κομισιόν για την αξιολόγηση. Τώρα, ε, προς τον κύριο Φανίστερόι έχω να κάνω ένα ερώτημα, γιατί δεν κατάλαβα καλά. Χθες, ε, δεν ξέρω αν το συζητήσατε, μιλάω για τις ε, μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Ε, προφανώς αυτή τη στιγμή ο εισηγητής του ελεκτικού συνεδρίου μίλησε για το κριτήριο αυτό και είπε ότι είναι ακατάλληλο. Υπάρχει πρόθεση να αναδιαπραγματευτείτε με την Κομισιόν το σημείο αυτό, την εισαγωγή δηλαδή αυτών των προϋποθέσεων στον γενικό κανονισμό των διαφόρων ταμείων. και ο εισηγητή, ο κύριος Μποστινάρου, ζητάει στη δική του έκθεση να αναθεωρηθεί αυτό το σημείο ε, για το Ταμείο Συνοχής. Λαμπέρ, θες να απαντήσεις, θες να αντιδράσεις και μετά θα ήθελα να ακούσουμε και τις αντιδράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Στο έγγραφο εργασίας μας υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία, μια σειρά από προβληματισμοί και προσανατολισμοί. Θέλω να ξεκινήσω με το, ταμείο, με το αποθεματικό απόδοσης. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Δεν τη βλέπουμε. Θα παρουσιάσουμε τροπολογίες. Έτσι. Ούτω ώστε αυτή η πρόταση να μην περάσει. Και θα, δώσω, και θα δούμε τι θα προκύψει, τι θα δώσει αυτό. Υπάρχει μια πλειοψηφία πάντως που δεν επιθυμεί αυτό το αποθεματικό. Αν σε περίοδους κρίσης θεωρούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί, ε, δεν πρέπει να το προωθήσουμε. Όταν διστάζουμε, δεν έχει νόημα να προωθήσουμε κάτι, γιατί αλλιώς θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά θα δημιουργήσει λύσεις. Αυτή είναι η στάση μα. Εάν μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε διευκρινήσεις μέσω τροπολογιών, τόσο το καλύτερο, αλλά δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε εδώ ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με περιτά στολίδια. Δεύτερον, ο μηχανισμός διασύνδεσης για την Ευρώπη, το Connecting Europe. Χθε είδαμε ότι οι δύο εισηγητές είναι σύμφωνοι ούτως ώστε ένα τμήμα των διαθέσιμων μέσων να περάσουν σε ένα άλλο πλαίσιο με μια κεντρική διαχείριση. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό το μέσο, σε αυτό το μηχανισμό. Έτσι το λέμε ξεκάθαρα. Τέθηκαν διάφορα ερωτήματα. Τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτό το σημείο και στην αρχή της συνοχής που διέπει το Ταμείο συνοχή και την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι ακόμα έτσι, ασαφή, αμφίσιμα. Θα πρέπει να θέσουμε ερωτήσεις επί του κανονισμού και ε, στα πλαίσια της νομοδότησης που θα εκπονήσει η Επιτροπή Μεταφορών. Και εκεί θα πρέπει να θέσουμε τροπολογίες. Όταν παίρνουμε και κοιτάμε τα project, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες. Και έχουμε την εντύπωση ότι ο κανόνας που ισχύει είναι όποιος έρθει πρώτος, αυτός βολεύεται, αυτός εξυπηρετείται. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να το διορθώσουμε. Θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα και για τα κριτήρια εφαρμογής της συνοχής, της αρχής της συνοχής πρέπει να υπάρχει μια καλή εδαφική κατανομή. Δεν μπορεί αυτό που φτάσει πρώτος να εξυπηρετείται καλύτερα και οι άλλοι να του ξεχνάμε. Αυτή πρέπει να είναι η στάση μα χωρί ε, αρνητικές στάσεις. Ε, τώρα, για το κάπινγκ, για το ανώτατο όριο. Μίλησα πάρα πολύ χθε. Ήταν ε, παρόν και ο πρόεδρο τη επιτροπή προπολογισμών. Και εκεί θα πρέπει να πάρουμε θέση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος ανισορροπίας Έχουμε ένα νότατο όριο. Έχουμε κάποια ποσοστά απορρόφησης. Έχουμε και κάποια κριτήρια για την ε, κινητοποίηση των ταμείων. Εντάξει. Καλώς. Τώρα, κάποια μέτρα, ε, κάποια κράτη έχουν πάρει ε, μέτρα αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν τακτοποιήσει τα δημοσιονομικά τους και παίρνουν λιγότερα από το ταμείο. Αυτό γύρει ερωτηματικά, δημιουργεί δυσκολίες. Στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τροπολογίες για να δώσουμε την δική μας γνώμη, αλλά και για να ζητήσουμε διευκρινήσεις. Τέλος, η αιρεσιμότητα. Το συζητήσαμε μαζί την περασμένη φορά. Θα γίνεται εκ των προτέρων, ε, εκ των, προτέρων, εκ υστέρων, εξάντε, εξ με βάση κριτήρια τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Όλα αυτά τα συζητήσαμε. Αυτό που είναι ανοιχτό ακόμα, που δεν έχει αποφασιστεί, είναι αν είμαστε αντίθετοι στην, ε, στις μακροοικονομικές προϋποθέσεις, μακροοικονομική αιρεσιμότητα, τι γίνεται με τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί στα πλαίσια του six-pack, του πακέτου των 6 μέτρων, των 6 νομοθετικών μέτρων, για την ε, χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται, πώς θα συγχωνεύσουμε, πώς θα συγκεράσουμε τη θέση μας ε, με τα όσα έχουμε αποφασίσει στα πλαίσια του six-pack. Το θέμα δεν έχει κλείσει λοιπόν. Θα πρέπει να υπρασπιστούμε τη θέση μας όπως την παρουσιάσαμε στο έγγραφο εργασία μα. μας. Υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Τα νέα μέσα. Τα νέα 4 ή 5 καινούργια μέσα που αφορούν την πολιτική υπέρ των πόλεων. Θα τα εξετάσουμε αυτά τα έγγραφα στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ. Τέλος. θα σας προσκαλέσουμε, ούτως ώστε να σκεφτούμε ομού ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα κείμενα. Τώρα, για τα τρία θέματα μπορείτε, Κομισιό, να απαντήσετε. πέντε λεφτά. Thank you. Um, για το κάπινγκ, την οροφή. Νομίζω ότι ο Νίκολας Μαρτιν έδωσε απάντηση χτες. Οπότε δεν θα επισέλθω. Ένα σχόλιο για την μακροοικονομική αρεσιμότητα, για την μακροαιρεσιμότητα μάλλον. Η συζήτηση έχει εστιαστεί πιο πολύ στις κυρώσεις ως τώρα και ο Νίκολας ε, χτες εξήγησε την φιλοσοφία. Το άρθρο 21 της πρότασης του, κανονισμού, του γενικού κανονισμού, του νέου γενικού κανονισμού, πηγαίνει πολύ πιο μακριά. Προτείνει μια προσέγγιση και προληπτική ε, και διορθωτική και προωθεί έναν διάλογο ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πριν ε, διονγκωθούν. Οπότε διαβάστε το άρθρο 21, όλο μαζί όμως, και όχι μόνο το κομμάτι που αφορά τις κυρώσεις. Τώρα, για το αποθεματικό απόδοσης ή επίδοσης. Νομίζουμε ότι δεν έχουν γίνει κατανοητές οι, προτάσει μα. μας. Δεν έχω χρόνο να σας εξηγήσω λεπτομερώ, αλλά να σα πω τι δεν είναι αυτό το απόθεμα. Πρώτον, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό απόθεμα. Είναι ένα απόθεμα σε επίπεδο κράτους μέλους. Εκεί δημιουργείται το απόθεμα. Δεύτερη παρανόηση ότι δήθεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα προγράμματα για τα κονδύλια. Όχι. Ο μηχανισμός προτείνει η Κομισιόν είναι ο εξή. Κάθε πρόγραμμα καθορίζει τους δικούς του στόχους και τους τρόπους με τους οποίους θα τους επιτύχει. Το απόθεμα και η εκταμίευσή του έχει σχέση με την επίτευξη αυτών των στόχων τα προγράμματα δεν ανταγωνίζονται μεταξύ του. Δεν ανταγωνίζονται οι φτωχοί με του πλούσιους. Έχει, το απόθεμα έχει σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε πρόγραμμα. Επίσης, δεν είναι μηχανισμός που επιδιώκει να τιμωρήσει κάποιο κράτος μέλος ή κάποιο πρόγραμμα. Είναι ένας μηχανισμός κίνητρο. Γιατί δεν είναι τιμωρία, γιατί δεν είναι ποινή, γιατί οι πόροι οι οποίοι δεν θα εκταμιευτούν για το α ή το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμη στο κράτος μέλος για να εκταμιευθούν σε άλλα προγράμματα που πηγαίνουν καλά. Τέλος, η περιπλοκότητα. Η διαδικασία την οποία έχουμε προβλέψει είναι απλή. Πραγματικά απλή και σχεδόν μηχανική και αυτόματη, τολμώ να πω. Τα προγράμματα θα αξιολογούν το αν έχουν πετύχει τους στόχους τους, αν τους έχουν πετύχει έχουν πρόσβαση στο ε, απόθεμα, αν όχι δεν έχουν. Ασφαλώς δημιουργείται το θέμα του πού θα δίδονται οι πόροι, αυτά τα κονδύλια, αλλά ο μηχανισμός είναι απλός. Τώρα, ε, το μέσον Connecting Europe. Το ερώτημα είναι το πώς θα λειτουργήσει υπέρ της συνοχής το μέσον συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι ένας ε, μηχανισμός που είναι προσανατολισμένος πιο πολύ στις ανάγκες ε, με ήμι ε, ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς. Στόχος είναι η ανάπτυξη των λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών της συνοχής. Μιλάμε για project τα οποία είναι δύσκολα διότι είναι project που συνδέουν χώρες μεταξύ τους. Οπότε προτείνουμε έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που είναι ο μηχανισμός του Connecting Europe. Και αυτό συνεπώς Πάγεται μεταφορά ποσόνα από το Ταμείο Συνοχή στον μηχανισμό του Connecting Europe, προκειμένου αυτό να έχει επαρκή χρηματοδότηση. Νομίζω ότι τα πράγματα μέχρι εκεί είναι σαφή. Το θέμα το οποίο είναι εκρεμές είναι σαφές πως είναι το πώς ε, θα ε, καταμεριστούν τα κονδύλια. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εθνικό, στο εθνικό καταμερισμό Έτσι έχουμε σκεφτεί το σύστημα. Νομίζω ότι αυτό ε, δίνει αρκετές εγγύσεις έτσι ώστε ε, τα κράτη ε, να έχουν επαρκή πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα ήθελα να ακούσετε την πρότασή μου γιατί μας μένουν λιγότερο από δύο ώρες για τέσσερις κανονισμούς. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για όλους τους κανονισμούς. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο από μισή ώρα για κάθε κανονισμό. Οπότε ε, σκεφτείτε πριν ζητήσετε το λόγο. Θα ζη... Αφού μιλήσει ο ε, εισηγητή κάθε φορά, θα λέω ποιο θέλει το λόγο θα... και θα κλείνει η λίστα των ομιλητών. Δεν θα προσθέτω άλλου αργότερα. Οπότε, ξεκινάμε με την ομοδότηση Μαρία Ερηγόγεν Πέρε για το Κοινωνικό Ταμείο. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο έτσι ώστε να δούμε πόσο χρόνο θα δώσουμε σε κάθε ομιλητή. Σκεφτείτε το, ο λόγος στη Μαρία εντωμεταξύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επικεντρώσω την ανάλυση του εγγράφου εργασία ε, σε αυτά που μας ενώνουν καταρχήν. Μετά θα μιλήσω ε, για τη σχέση με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και μετά θα μιλήσω για το κοινωνικό ταμείο. Ε, ξεκινάμε από τον εξή κοινό παρανομαστή. Τρία σημεία. Πρώτον, σημασία τη προσθέμενη αξία του κοινωνικού ταμείου για την καταπολέμηση τη ανεργία, ε, υπέρ τη μείωση των ανισοτήτων, της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότητας και της ε, ισότητας στην κατάρτιση. Επίσης η ανάγκη να εξασφαλίσουμε την ελαστικότητα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και η ανάγκη της μείωσης του διοικητικού άχθους και της απλοποίησης με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα ταμεία. Τρίτον, η πρόθεση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και των και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων καθώς επίσης και των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τώρα, θέλω να εστιαστώ σε δύο θέματα τα οποία εξαρτώνται από τη γενική νομοθεσία αλλά έχουν σχέση και επηρεάζουν το κοινωνικό ταμείο. Πρώτον, η σημασία να ε, συνδυάσουμε την επαρκή χρηματοδότηση με το κοινωνικό ταμείο έτσι ώστε να του επιτρέψει αυτή να επιτύχει τους στόχους του αλλά ταυτόχρονα να δώσουν και στα κράτη-μέλη επαρκή ελαστικότητα στην κατανομή των ποσών των κονδυλίων σύμφωνα με τα όσα έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο θέμα, η σημερινή τροφικού προγράμματος 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου. Δεν είναι η πιο ιδανική λύση, αλλά είναι απαραίτητη για να μειώσουμε τη φτώχεια. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό και εξαρτώνται από αυτό εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε. Τώρα, πιο συγκεκριμένα θέματα για το Κοινωνικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά την αποστολή του και το πεδίο εφαρμογή, το άρθρο 2 και άρθρο 3 του Ταμείου, προτείνω κάποιε τροπολογίε πολύ συγκεκριμένε που θεωρώ απαραίτητε. Δηλαδή, αυτέ που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόληση με συγκεκριμένε ομάδε του πληθυσμού και τι ε, πολιτικέ ισότητας. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τι προτεραιότητες με αναφορά, με συμπερίληψη των μεταναστών, συγγνώμη, και με την προσαρμοσμένη κατάρτιση μεταξύ άλλων. Άρθρο 4. Θεματική συγκέντρωση και λογική συνοχή. Η Κομισιόν ε, καθιστά υποχρεωτική την συγκέντρωση χρηματοδότηση σε τέσσερι το πολύ άξονες σε περιφερειακό επίπεδο με ποσοστά 60, 40 και 80%. Σε εθνικό επίπεδο το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εγγυάται τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησης ε, για την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Επιμένω ότι αυτή η κατανομή είναι απολύτως απαραίτητη αυτό το 20% ιδιαίτερα, δεδομένου ότι πάνω από 113 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη ε, διατρέχουν τον κίνδυνο της κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Η συγκέντρωση σε τέσσερις μόνο προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο και με τόσο ψηλά ποσοστά μειώνει σαφέστατα πάρα πολύ την ευελιξία και την δυνατότητα να προσαρμόζονται οι παρεμβάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στι ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Συνεπώς, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του Ταμείου χρειάζεται η συγκέντρωση να γίνει με μικρότερα ποσοστά και οι προτεραιότητες επένδυσης να αυξηθούν στο αριθμό. Άρθρο 6. Συμμετοχή των εταίρων. Η Κομισιόν προτείνει την αυξημένη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων και την ε, πρόσβασή τους σε χρηματοδοτούμενα μέτρα. Αυτό αυτό θα ήταν επαρκές για την συμμετοχή των μικρών ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλλά ε, χρειάζεται και η συμμετοχή των τοπικών και ψηφιακών ε, φορέων και αρχών γιατί δεν έχουν όλες τα ίδια μέσα και ικανότητες για παράδειγμα ε, στις ζώνες της υπαίθρου η, αρχή της ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών άρθρο 7 αυτό θα πρέπει να, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουν και τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα εμπόδια επίσης στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία και την σημασία να συμπεριλάβουμε επιδόματα και βοήθεια για τα εξαρτώμενα άτομα, παιδικούς σταθμούς, βρεφονικούς σταθμούς κλπ. Ε, πρόθεση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκριση άρθρο 8, εκεί είναι σημαντικό να αναφέρουμε την πραγματικότητα αυτών που υφίστανται διακρίσεις. Άρθρο 9, κοινωνική καινοτομία, βασική καινοτομία αυτή της πρότασης. Αυτή η συμπερίληψη θα μπορούσε να βελτιωθεί αν ορίσουμε ε, σχέση με τις ε, ποινές ε, των γενικών γραμμών και των περισσιακών προγραμμάτων έτσι ώστε να αποφύγουμε αποκομμένα και κατακαιρματισμένα μέτρα. Στη διεθνική συνεργασία άρθρο 10 Χρειάζεται να εισάγουμε επίσης και την διαπεριφερειακή συνασία και να επιμείνουμε για την ανάγκη τεχνικής συνδρομής και συνοχής ανάμεσα σε διεθνικά θέματα και τους ε, θεματικούς στόχους για να εγγυηθούμε την ε, επιτυχία μακροπρόθεσμα. Από την άλλη μεριά, η κατάρτιση των καταλόγων, των θεματικών καταλόγων είναι πολύ περιοριστική και αφήνει εκτός νυμφώνος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήταν χρήσιμο ο κατάλογο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να επιτρέψουμε έτσι τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο, να δώσουμε δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του. Ε, ε, ιδιαιτερότητε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες, άρθρο 12. Ο καινούργιο κανονισμό προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στρατηγικέ ε, τοπικής ανάπτυξης. Πολύ καλό δείχνει αυτό, δεδομένη τη ανάγκη να εστιάσουμε ε, ε, δεδομένου τη εστίαση της πόλης ε, της πολιτικής συνοχής. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διάσταση πέθρου στις εδαφικές ιδιαιτερότητε. άρθρο 14. απλοποιημένα κόστη. αυτό απλοποιεί πράγματι τη λειτουργία του συστήματος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευελιξία στην υλοποίηση των προγραμμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού άχθους με στόχο να ενδυναμώσουμε και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των δικαιωχών. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ορισμένες διευκρινήσεις στον ορισμό των βασικών ε, ενιών και της εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Οι κοινοί δείκτες υλοποίησης, εκτέλεσης ε, προβλέπονται από την Κομισιόν ε, για να μετρηθούν τα αποτέλεσματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτοί οι δείκτες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ε, συμμετέχοντες και φορείς. Σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δίδονται από τους συμμετέχοντες υπάρχουν κοινοί δείκτες. Με στόχο να έχουμε με περισσότερο πιο λεπτομερή εικόνα των επενδύσεων του Κοινωνικού Ταμείου και να μετρήσουμε τον αντίκτυπο του αναφύλου, χρειάζεται οι δείκτες να είναι πιο λεπτομερείς, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν και την πτυχή του φύλου. Πέραν από την άλλη μεριά τη συμπερίληψη των ε, ορισμένων δικτών, μα πιο μακροπρόθεσμων, ορισμένοι πρόσθετοι δείκτες θα είναι χρήσιμοι, ορισμένοι δείκτες αντικτύπου θα ήταν ε, πιο χρήσιμοι. Όπως σας έλεγα και στην αρχή της ε, παρουσίασής μου, ε, η τροποποίηση οι τροποποίησεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 2 Μαΐου και θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση 21 Μαΐου. 1,5 μήνα πριν την υιοθέτηση ε, της ε, ε, έκθεσης. Ε, οπότε στην Ολομέλεια. Οπότε ελπίζω να μας βοηθήσετε. Ευχαριστούμε Μαρία. Τρεις ομιλητές έχω. Κλείνω τον κατάλογο. Better. Uh, so I hope three minutes will be sufficient for all of you. Uh, Τρία λεφτά όλοι μαζί. Κυρία Λουκατσένσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, κυρία Συγήτρια. Άκουσα όλες τις ε, παρατηρήσεις ε, που έκανε, όλα τα σχόλιά της. Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε. μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες ε, στις διάφορες πτυχές του κοινωνικού ταμείου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση το κοινωνικό ταμείο είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο για να καταπολεμήσουμε τα ανεργία, τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών, την καταπολέμηση της φτώχειας και την καλύτερη κοινωνική ένταξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το ταμείο Και οι διατάξει που υπάρχουν στην έκθεση είναι πολύ σημαντικέ. Το μόνο που χρειάζεται ίσω είναι λίγο περισσότερη ευελιξία. Άλλο σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ring fencing. Δηλαδή, το πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προτάσεις που γίνονται δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες μεταξύ περιφερειών και των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν ειδικέ ανάγκες από ορισμένε τοπικές αρχές και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό στα πλαίσια του προγραμματισμού. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να σκεφτούμε να βρούμε πιο ευέλικτες λύσεις. Κάτι άλλο η ισότητα ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά. Και εδώ συχνά μιλάμε για τις διαφορές αυτές και εδώ και στην Ολομέλεια για τις διαφορές ε, τις μισθολογικές. Συχνά έχουμε και διατάξεις σε διάφορα νομοθετικά κείμενα, αλλά αυτά μοιάζουν να είναι απλά λόγια. Μοιάζει σαν να μην εποφελούνται καθόλου οι γυναίκες. Ξέρω πολύ καλά ότι οι μισθολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών είναι περίπου 20%. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο της ανισότητας. Θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια, ούτω ώστε να επιτρέψουμε στην, στις γυναίκες να επανέλθουν στην αγορά εργασίας όταν γεννήσουν, Φερρυπίν. Η απασχόληση των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές γυναίκες σήμερα δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα μπορεί να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους σήμερα, επειδή υπάρχουν πολλές ε, συρρυκνώσεις, πολλές απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Επίσης υπάρχει και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ίσως θα πρέπει να συνδυάσουμε τους στόχους του Κοινωνικού Ταμείου με τους στόχους του Ταμείου Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους ε, εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους μετά από μαζικές απολύσεις, που είναι συνέπεια αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης. Ε, η κρίση έδωσε σήμερα στο κοινωνικό ταμείο ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Γίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ταμείο, ούτω ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι μαζί με τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο οικονομικό κύκλο και στις απαιτήσει της αγοράς. Υπάρχει και ένα θέμα εκπαίδευσης επίσης. Θα πρέπει ο καθένας ε, να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, να μπορεί να μαθαίνει διαβίου. Νομίζω ότι το κείμενο μου θα πρέπει να μπει περισσότερο σε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες, ούτω ώστε να δούμε τι είδους ε, κατάρτιση μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί, τι είδους ε, κατάρτιση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το κοινωνικό ταμείο. Επίσης, σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέμε ότι πρέπει να αυξήσουμε την ηλικία σταξιοδότησης. Ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε είναι ότι ο πληθυσμό γυράσκει, υπάρχει ένα ποσοστό γεννήσεων πολύ χαμηλό, όλο και πιο χαμηλό, άρα πρέπει να δουλεύουμε πιο πολύ. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα άτομα ε, πάνω από 50 ας πούμε, που χάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς θα εξασφαλίσουμε την ενεργή γύρανση του πληθυσμού. Τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε ε, οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι να κρατάνε τη δουλειά τους μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Θέλω να πω και κάτι που μου αρέσει να το λέω συχνά. Η κατάρτιση, κατάρτιση των εργαζομένων, ούτω ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας, στις νέες προσδοκίες των επιχειρήσεων. Ε, υπάρχουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που ε, δαπανώνται με τρόπο καθόλου αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά κατάρτιση συχνά. Ε, συχνά, ας πούμε, δαπανάμε τα λεφτά του Κοινωνικού Ταμείου γιατί πρέπει να δαπανηθούν. Αν όμως θέλουμε και την αποτελεσματικότητα ε, μετά από τις δαπάνες ε, των ε, κονδυλίων, βλέπουμε ότι συχνά ξοδεύονται χρήματα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπω ότι άτομα περνάνε από μια διαδικασία κατάρτισης και δεν είναι παρόλα αυτά πιο ελκυστικά για την αγορά εργασίας. Πώς μπορούμε να ξοδεύουμε κάποια λεφτά ούτως ώστε το άτομο να επανέρχεται στην αγορά εργασίας και να βρίσκει μια νέα θέση απασχόλησης. Ε, το ρώτησα αυτό και στον Επίτροπο. Και το ρώτησα ποια είναι τα αποτελέσματα των δαπανών που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Δηλαδή, ποια, τι ποσοστό από τα άτομα τα οποία ακολούθησαν μια κατάρτιση μπορούσαν να βρουν μια νέα απασχόληση. Έχω θέσει αυτά τα ερωτήματα, όπως σας είπα. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης και την αρχή νήσιν 3. Είχαμε το νήσιν αλλά σήμερα θα πρέπει να έχουμε και κονδύλια τα οποία ξοδεύονται πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και μας δίνουν μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία κατά την υλοποίηση των σχεδίων. Πρέπει επίσης να διευκρινιστούν και άλλα σημεία. Κάποιοι ορισμοί φερρυπίν και οι προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Η συγγήτρια έχει δίκιο ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί πριν ε, καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά χάρη στις τροπολογίες που θα καταθέσουμε θα μπορέσουμε να επιφέρουμε και τροποποίηση το κείμενο. Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να σέβεστε τα τρία λεφτά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα θέματα που θέλουμε σήμερα. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρωτοβουλία να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί το, τελευταίο πλαίσιο που είχαμε δεν ήταν το πιο αποτελεσματικό. Όταν μιλάμε για δείκτες και για την εφαρμογή για τους διάφορους κοινωνικούς τομείς, ε, σας εφιστώ την προσοχή στους δείκτες που θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ε, στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Οι δείκτες αφορούν τους διάφορους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες. Οι ανάγκες της κάθε χώρας δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτως ώστε να δαπαντώνται με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο τα χρήματα. Η αγορά εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη από τους δείχτες. Τώρα περνάμε μέσα από αλλαγές, τις ονομάζουμε μεταρρυθμίσεις, ιδίως στα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα νέα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις οικονομίες μας και την αγορά εργασίας μας στα δυτικά πρότυπα. Και υποστηρίζω αυτό που είπε η συνάδελφος, ότι οι προτάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Θα έπρεπε να το κάνουν όμως αυτό. Επομένως, οι επόμενες προτάσεις και το επόμενο πλαίσιο θα πρέπει να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει ε, στα μελη θα, πρέπει, μάλλον να έρθουμε σε επαφή με τις ε, εθνικές αρχές και με τις περιφερειακές αρχές. Α, μερικές φορές οι περιφέρειες απλώς υφίστανται, απλώς είναι ε, υποχρεωμένες να δεχτούν αυτά που τους επιβάλλουμε. Ε, αν ας πούμε μία περιφέρεια ε, έχει δυναμικό σε ένα συγκεκριμένο τομέα, δεν πρέπει να την εξαναγκάζουμε να ασχοληθεί με ένα τελείως διαφορετικό τομέα, μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν λεφτά διαθέσιμα για τον άλλο τομέα. Ε, γιατί αυτό θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, αυτή η προσαρμογή. Θα πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση α, συγχρηματοδότησης. Και θέλω να προτείνω ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησεων για την συγχρηματοδότηση το τονίζω, συγχρηματοδότηση. Και στο τέλος κάθε έτους θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους κινδύνους, ούτω ώστε αυτό το ταμείο και τα λεφτά που πηγαίνουν στο Ταμείο Εγγυήσεων να μπορούν να χρησιμοποιούνται την επόμενη χρονιά. Το Ταμείο δεν θα χάνει τίποτα, αλλά θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεργάζεται με τις εθνικές τράπεζες και οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στη συγχρηματοδότηση μέσω αυτού του Ταμείου Εγγύσεων. Θα είναι ένα τεράστιο βήμα αυτό. Θα μπορέσουμε δηλαδή να ε, απελευθερώσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να φτάσουν τελικά στους δικαιούχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει χρήματα για την υποστήριξη τομεακών πολιτικών. Και θα πρέπει τα χρήματα αυτά ε, να συνάδουν με την ευρωπαϊκή στρατηγική ή τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Τέλος, υπάρχει το εθνικό διοικητικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ την προσοχή σε αυτό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει προτάσεις σε σχέση με αυτό το εθνικό διοικητικό πλαίσιο που θα πρέπει να συμφωνηθεί πριν υπογραφεί η συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δαπανώνται τα δημόσια χρήματα. Ποια είναι η αρχή διαχείρισης, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποια είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων κτλ. Μιλάω για όλα αυτά τα θέματα. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, με την οποία έχω και άμεσα συνεργαστεί. Το θέμα προχωράει πολύ καλά. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς ε, τομείς συνένεσης. Δεύτερον, ε, εγώ δεν ξέρω τι πρότεινα προαλήσαν για το Ταμείο, γιατί εδώ έχουμε άτομα που δεν έχουν χρήματα δικά τους και θα χρειαστούν δημόσια χρήματα. Και το θέμα είναι κατά πόσον τα κράτη-μέλη θέλουν να εξαλείψουν τη φτώχεια και την ανεργία και κατά πόσον γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουν χρήματα ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Αλλά είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί από τέτοια τα κράτη-μέλη. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στον συγκεκριμένο ε, κανονισμό του Ταμείου και σε αυτά που είπε η εξηγητής. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει διαβρινθεί ε, ο κανονισμός επένδυσης, γι' αυτό ο κανονισμός έχει πολλά χρήματα ε, στη διάθεσή του το Ταμείο. Εμείς υποστηρίζουμε και τα, τους δύο νέους τομείς που είναι συμφωνούν και με την στρατηγική της Ευρώπης 2020. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Βλέπω όμως στο συγκεκριμένο κείμενο ένα πρόβλημα. Γιατί δεν αντικατοπτρίζεται ο στόχος της φτώχειας όταν εξετάζουμε ε, ποιος είναι ο δικαιούχο τελικά. Γιατί διευρύνεται ο κανονισμός, διευρύνονται τα χρήματα και διευρύνεται άρα και η ομάδα των δικαιούχων Χωρί να του ορίζουμε με σαφήνεια. Επίσης το άρθρο 4 είναι για μας προβληματικό. Ακόμα και αν κεντρώσουμε τους πόρους και θα είχε νόημα κάτι τέτοιο, δεν θα λειτουργήσει. Ας πούμε, φτώχεια. Ένα κράτος μέλος συγκεντρώνει τους μεγάλους πόρους του ταμείου, του κοινωνικού ταμείου, για ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της ένδυας. Πλήρες. Αλλά με εξετάσουμε τις λεπτομέρειες θα δούμε ότι υπάρχουν 7 συγκεκριμένα θέματα που τίθενται εδώ για την πραγματοποίηση του προγράμματος κατά της ένδυας. Και θα πρέπει ίσως για να καταπολεμήσω τη φτώχεια να έχω και κάποιες προτεραιότητες στον τομέα της απασχόλησης. Έχω ήδη εννέα δηλαδή προτεραιότητες ακόμα και αν ε, είμαι πολύ συγκεκριμένη για το θέμα της ε, ένθειας. Δεν θα λειτουργήσει λοιπόν. Δηλαδή καλή είναι η βάση αλλά η διατύπωση με τα ε, τέσσερα αυτά δεν είναι σωστή. Και μπορούσα να πω θα πάρω τα θεματικά κύρια θέματα και στο τον συνδυασμό τους για να πετύχω το 1 ως 11 στον γενικό κανονισμό. Και να πω στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τόσο από το ε, κοινωνικό ταμείο. Εντάξει αυτό. Αλλά αν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, θα έλεγα, α πούμε το καλύτερο παράδειγμα είναι ένα καλό πρόγραμμα για τη φτώχεια, ένα καλό πρόγραμμα για την παιδεία, θα πρέπει να έχω περισσότερε δυνατότητε συνδυασμού και να είμαι συγκεντρωμένη παρόλα αυτά στο αποτέλεσμα. Ένα αυτό. Θα πρέπει να συζητηθεί. Γιατί κατά γνώμη μου δεν ε, λειτουργεί όπως θα έπρεπε και δεν θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα της μείωσης ε, της φτώχειας, τη μείωση των, ε, του αριθμού των παιδιών που διακόπτουν το σχολείο, τη μείωση των ατόμων που απειλούνται από μακροχρόνια ανεργία. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το άρθρο 6 για τις εταιρικές σχέσεις, όπου γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων των κρατών μελών που είναι καλύτερα ανεπτυγμένε και τι άλλε. Ε, δεν θέλω όμω εγώ μια τέτοια μείωση γιατί σε όλε τι χώρε μέλη, ακόμη και στι πλούσιες, υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων για να εμπλακούν εδώ, για να παίξουν εδώ, εδώ τι χρειαζόμαστε πάντου. Όσον αφορά λοιπόν τα δύο, το 2 και το 3 θα πρέπει να ισχύει για όλους. Χαίρομαι που η εισηγήτρια αποφάσισε να βρει αυτή τη λύση για το επιστηστικό πρόγραμμα. Και εμείς το συζητήσαμε το διαμακρόν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε, εντάξει, με το επιστηστικό πρόγραμμα έχουμε καλύψει το, την φτώχεια του 20% και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό είναι μεγάλη κίνδυνο εάν ακολουθούσαμε αυτό που είχε προτείνει η εισηγήτρια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εν ώψη της σφαιρικής κατάστασης που έχουμε για τα έξι αυτά κράτη-μέλη, έξι έχουμε εδώ, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και περνάμε πάλι στο άρθρο 4 όπου έχουμε το θέμα της συγκέντρωσης. Αν ανοίγαμε λίγο τη συγκέντρωση αυτή, αν μπορούμε δηλαδή να έχουμε περισσότερα θέματα για να πετύχουμε ένα θεματικό στόχο, θα υπήρχε δυνατότητα συνδυασμού μεταξύ του πιστιστικού προγράμματος και ενό άλλου προγράμματος. Για τα σε έξι αυτέ χώρες κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία άλλη λύση και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό έτσι. Γιατί είναι καλό νομίζω για την επίτευξη των Έχουμε ένα συνδυασμό με το πρόγραμμα της καταπολέμησης της ένδυας. Ε, θα μπορέσουμε νομίζω έτσι καλά να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι καλό γιατί τις λόγω έξι χώρες μέλη. Ε, στηρίζω την ε, ε ησυχήτρια όσον αφορά την ε, παράγραφη για την προστασία. Έχω ένα πρόβλημα που δεν ξέρω. Η κυρία Μπέρκοβιτς είναι εδώ, δεν ξέρω αν μπορεί να μου απαντήσει. Γιατί κάτι που δεν υπάρχει ίσως στο κοινωνικό ταμείο, στην κανονισμό για το κοινωνικό ταμείο. Τουλάχιστον δεν το βρήκα πουθενά. Στην ομάδα εργασία είχαμε συζητήσει για εκείνα τα σχέδια, τα μικρά, που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτής της προκαταρτικής χρηματοδότησης, να υπάρχει μεγαλύτερη προχρηματοδότηση από την Κομισιόν, ούτω ώστε το κίνδυνο να μην ε, τον, τον κίνδυνο να μην τον επομιστούν οι δικαιούχοι. Δηλαδή, εν τελευταία αναλύση όλο το βάρο της προχρηματοδότηση να μην παραμείνει σε εκείνου που έχουν υποβάλει τα σχέδια αυτά δεν βρήκα εγώ που υπάρχει κάποια αλλαγή ότι η Κομισιό δηλαδή χρηματοδοτεί καταρχήν με υψηλότερο ποσοστό ένα πρόγραμμα στην αρχή και στο τέλος με χαμηλότερο ποσοστό. Έτσι ούτω ώστε οι μικρές ομάδες πραγματικά καταρχήν να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Και να μην λένε ότι εντάξει δεν μπορούμε να υπομισθούν αυτό τον οικονομικό κίνδυνο. Βοηθήστε με να το βρω, εγώ δεν το βρήκα πουθενά. Δύο λεφτά παρακαλώ, το πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες σας για τις παρατηρήσεις σας. Όλοι ξέρουμε και είμαστε σίγουροι πως θα συνεργαστούμε έτσι ώστε η έκθεση να είναι όσο πιο στέρεη γίνεται. Γιατί θέλουμε αυτό το ταμείο να είναι ισχυρό ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Ε, ζητάτε να είναι το ταμείο αυτό πιο ευέλικτο, να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων, πραγματική υποστήριξη για τους, ανέργους, για ανέργους και ιδιαίτερος για τους νέους προσαρμογή της παιδείας και της κατάρτισης, ε, εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αγορά εργασία και να είναι ένα μέσο συγχρηματοδότησης. Ε, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για να προσπαθήσουμε αυτή η έκθεση πραγματικά να είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει να απαντήσει η Κομισιόν στο σύντομα, ίσως. Μάλιστα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα της Ελίζαβετ Σρέντερ όσον αφορά την προγραμματιδότηση των μικρών σχεδίων. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό για την προχρηματοδότηση. Παρόλο όμως, αυτό που κάνει είναι ότι αλλάζει τον χρηματοδοτικό μηχανισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν έχει σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Και αυτό το έχουμε στο άρθρο 121 γάμα. Γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στο κράτος μόνος μόνο εάν μπορεί το κράτος να αποδείξει ότι έχουν δοθεί τα χρήματα στο δικαιούχο. Εν αντιθέσει προς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ένα στοιχείο αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι η προχρηματοδότηση που προβλέπεται που επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να έχει πάντα αρκετή ε, ρευστότητα. Αυτά τα δύο από κοινού πετυχαίνουν αυτό που προτείνεται ακριβώς. Ότι επιτρέπεται δηλαδή στα κράτη-μέλη να προχρηματοδοτήσουν μικρά σχέδια. Αυτή είναι η τεχνική ερώτηση στο, απάντηση στο ερώτημα σας και θα δώσω το λόγο στο Τόμας Πέντενη για να απαντήσει τα άλλα ερωτήματα. Ναι, πράγματι υπήρχαν πολλές ερωτήσει Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δεν μπορώ να καλύψω όλα, να καλύψω όλα τα σημεία. Το ένα αφορούσε το θέμα της ε, συγκέντρωσης ε, σε σχέση με την ευελιξία. Νομίζω ότι η πρόταση προβλέπει και τα δύο, γιατί δεν λέγεται ακριβώς ποιες ε, περιφέρειες και ποιε προτεραιότητες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από το κράτημα. Λέει ότι έχετε την επιλογή από 10 8 μέσα σε τέσσερα θέματα. Και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες στα πιο επίγοντα θέματα. Και έχουμε διαφορετικό ποσοστό πρότασης για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν κάποιους άλλους τομείς που δεν εντάσσονται ακριβώς στους τέσσερις τομεί που προβλέπει ο κανονισμός για το Ταμείο. Όσον αφορά το θέμα, του δείκτες και την αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε ε, ένα σχέδιο προετοιμάσει για τον κανονισμό αυτό όσον αφορά τις επιπτώσεις του, την αποτελεσματική χρήση των πόρων για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα προτείνουμε αυτούς τους κοινού ε, δείκτες και όσον αφορά την απόδοση αλλά και για το Ταμείο όσον αφορά το θέμα των αποτελεσμάτων. Αυτά όλα θα συμπληρωθούν από προγράμματα και προτεραιότητες συγκεκριμένων δικτών που θα παρακολουθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για πολύ πολύ καθορισμένα σχέδια. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις, η Κομισιόν στην πρότασή της έχει προβλέψει οι αρχές των κρατών μελών να συλλέγουν στοιχεία συμμετεχόνων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά διάρκεια προόδου των προγραμμάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία από κοινού θα μας δώσουν περισσότερα, θα μας εξοπλίσουν καλύτερα, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σημείωσα επίσης τις αναφορές που γίνονται για την χρηματοδότηση. Ναι, ακούσαμε προσεκτικά το Κοινοβούλιο που λέει ότι είναι κατά των εθνικών ε, συμβολών ή των εθνικών ορίων για το Ταμείο. Η πρώτη Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα ποσοστά ανακατηγορία περιφέρειας σε ένα κράτος μέλος αυτά τα ελάχιστα ποσοστά είναι προσαρμοσμένα στην ιστορική εικόνα που έχουμε για τις εν λόγω περιφέρειες. Όσον αφορά το θέμα του φύλου και της πολλαπλής διάκρισης, νομίζω ότι ο κανονισμός επιτρέπει αρκετή ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό τομέα και τα εν λόγω προβλήματα. Γιατί το θέμα του να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φίλων δεν θα εξεταστεί ξεχωριστά. Χρειαζόνται πολλά συνοδευτικά μέτρα που υιοθετούν οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σωστή νομική βάση για να μπορέσει να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες. Όσον αφορά τις πολλαπλές διακρίσεις, θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό γενικών διατάξεων που απαιτεί από τα κράτη-μέλη τον καθορισμό των στρατηγικών τους για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλή ε, διάκριση και που βρίσκονται ήδη μέσα σε πλαίσια σχέσεις, ε, ε, εταιρικής σχέσης αν θέλετε και αυτό δεν είναι θέμα μόνο του κοινωνικού ταμείου αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνδυάσουν τα διάφορα ταμεία που έχουν στη διάθεσή του. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε η κυρία Σρότερ, ένα θέμα σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις και τα ποσά που προβλέπονται για τους κοινωνικούς εταίρους και τους μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ακριβώς για τους κοινωνικούς εταίρους έχουμε αυτούς τις ε, διατάξεις ε, σήμερα και δεν θεωρήσαμε ότι πρέπει να αλλάξουν γιατί στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή πιο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη τα ε, χρήματα ε, είναι επαρκή που διατίθενται. Δεν βλέπουμε να υπάρχει εδώ μια πρόκληση που θα πρέπει να επιλύσουμε συμπληρωματικά. Επίσης αυτό που εισαγάγουμε είναι μια υποχρεώση για τα κράτη-μέλη να έχουν παρόμοια προσέγγιση στο στη, ε, δημιουργία των δυνατοτήτων του μη κυβερνικού τομέα. Σημειώσαμε επίσης αυτό που είπατε για το επιστηστικό ε, πρόγραμμα και ο Επίτροπος μου και ο Επίτροπος Σολωστή περισσότερη φορά στο Ρασβούργο έκανα τα απαραίτητα σχόλια και η Κομισιόν θα φροντίσει να είναι σωστή η πρωτοβουλία που υποβάλλει στο μέλλον. Όσον αφορά το θέμα της προχρηματοδότησης για τα μικρά προγράμματα, τα οποία είπε ότι έπρεπε να ελεγχθεί. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το κανονισμός για το κοινωνικό ταμείο. Προβλέπει συγκεκριμένε διατάξει που καθιστούν υποχρεωτικό οι διοικητικέ αρχέ να έχουν προβλέψει συγκεκριμένα ε, κονδύλια για τα μικρά αυτά σχέδια με ένα μέγιστο ποσό 50.000 ευρώ και νομίζω ότι για όλα αυτά τα μικρά ε, προγράμματα και σχέδια θα μπορέσει η διάταξη αυτή να επιτρέψει την πολύ πιο γλίγορη πρόσβαση στα, στη χρηματοδότηση. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω χρόνο, Πρόεδρε. Αλλιώ θα σα είχα σταματήσει εγώ. Ευχαριστώ που σταματήσατε. Ευχαριστούμε για τι εξηγήσει. Έχουμε 45 λεπτά για τρει κανονισμού πια. Οι 25 λεπτά θα αφιερώσουν στον πρώτο κανονισμό σε κάθε κανονισμό. Ε, και στα 25 λεπτά σταματάμε. Ε, εδαφική συνεργασία. Ποιο θέλει το λόγο μετά την ε, εισηγήτρια, ε, τη Ρίκα Μάνερ. Ευχαριστώ, Ρίκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συντάσσω και εγώ το έγγραφο εργασία μου. Σας ε, έχω αποστείλει ένα αντίγραφο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το έχετε διαβάσει λοιπόν φαντάζομαι. Επτά είναι τα θέματα στα οποία θα εστιαστούμε. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη για αυτές τις ερωτήσεις, για αυτά τα θέματα. Είναι αυτά που πιο πολύ, όπως σας είπα, θα μας απασχολήσουν τον κανονισμό εδαφικής συνεργασίας. Καταρχήν σας πω το εξής. Πρέπει να εξασφάλισουμε καλύτερη ευκρίνεια του ρόλου που μπορεί να παίξει το Ταμείο Προφερειακής Ανάπτυξης ε, πιο πολύ από το παρελθόν. Πρέπει να είμαστε σαφείς, να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλπ. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, θέμα της χρηματοδότησης. Δημοσιονομικό θέμα. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το κοινοβούλιο θα το συζητήσει. Ιδιαίτερα θα συζητήσει τα θέματα τα σχετιζόμενα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρόσφατα υιοθετήσαμε μια έκθεση που συνδέεται στενά με την εδαφική συνεργασία. Και εκεί λέμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον το 80% του προπολογισμού. Η Κομισιόν μας υπέβαλε ένα ε, ποσό 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει 3,8 ε, 3,48% του συνολικού προπολογισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αδέρφους αν ε, θα επιμείνουν στις δικές, στη δική μας άποψη αυτό που είχαμε προτείνει δηλαδή το 7% γιατί μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να φτάσουμε στο 7%. Μετά, ευελιξία. Στην προηγούμενη, περίοδο, στην προηγούμενη περίοδο μπορούσαμε να μεταφέρουμε ποσά ε, ανάμεσα στα κεφάλαια α, β και γ, ανάλογα με τι ανάγκε. Για παράδειγμα, να αφιερώσουμε μεγαλύτερα κονδύλια στην ε, διασυνορική συνεργασία όταν το χρειαζόμασταν. Τώρα, με την καινούργια πρόταση τη Κομισιόν, δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρίμα που εγκαταλείπεται αυτή η ευελιξία. Θα Θέλαμε βέβαια η Κομισιόν να σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότηση αυτή η ευελιξία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, προβλέπεται το 75% τη συγχρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. Ε, το θέμα θα συνεχίσει να συζητείτε. Για όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ισχύει το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότηση για την απλοποίηση του πρόγραμματος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ήθελα να μου πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε. Μετά η Κομισιόν προτείνει ένα 6% για τεχνική ενίσχυση στην υλοποίηση. Καλό αυτό. Το ερώτημα είναι αν χρειάζεται κάτι ψηλότερο. Τώρα, για τη σύνδεση με άλλα προγράμματα. Το έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει μια σύνδεση ανάμεσα στα προγράμματα Εδαφική συνεργασία με τα άλλα προγράμματα, γιατί γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας ε, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να λειτουργήσουν καλύτερα. Θα ήθελα να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα και θα ήθελα επίσης η Κομισιόν να μας κάνει προτάσει, πιο σαφεί προτάσεις, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα και την συνέργειά τους. Τώρα, θεματική στόχη. Έχουμε ένα ολόκληρο κατάλογο με θεματικούς στόχους για τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Θα πρέπει να επιλεγούν τέσσερα, τέσσερις στόχοι. Αυτό για μένα δημιουργεί προβλήματα. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας είναι πολύ διαφορετικά από τα παραδοσιακά προγράμματα. Οπότε έχω την εντύπωση ότι οι τέσσερις ε, θεματικοί στόχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν ικανοποιούν τις ανάγκες. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Μια δυνατότητα θα ήταν να επιλέγονται τρεις ε, θεματικές προτεραιότητες και μετά οι περιφέρειες να μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες. Τώρα, οι διασυνοριακές μεταφορές. Χρειάζεται συνεργασία εδώ οπωσδήποτε και η Κομισιόν έχει πει ότι υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίηση αυτού, αυτών των προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων για τις υποδομές. Χρειάζομαστε όμως πιο σαφείς πληροφορίες από την Κομισιόν για αυτό το ζήτημα. Γιατί οι μεταφορές είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Μετά υπάρχει το θέμα της γύρανσης. Ίσως πρέπει να ε, συνδέσουμε και αυτό το ζήτημα με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Τώρα για τις μακροπεριφέρειες. Η συμφωνία αυτή, οι συμφωνίες αυτές ε, ε, αποτελούν πλέον τμήμα των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. Στο κεφάλαιο Β οι μακροπεριφέρειες έχουν ξεκινήσει, αποτελούν ένα θεματικό στόχο που μπορεί να επιλεγεί. Ο, ρόλος τους είναι ισορροπημένος στο κείμενο, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Απλοποίηση. η Κομισιόν μας έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης με μία αρχή διαχείριση μία διαχειριστική αρχή. Είναι πολύ καλό σημείο φετηρία. Και επί αυτού νομίζω συμφωνούμε όλοι. Κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν ε, ε, για την ευελιξία, κατά την άποψή μου πιστεύω ότι είναι αβαλιξία γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, με τον τρόπο που το θέλει. Αν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να υιοθετήσει αυτό το μηχανισμό, δεν είναι υποχρεωμένο. κάτι άλλο σχετικό με την απλοποίηση. Υπάρχει το 15% για ε, για, τα, για το κόστος ε, του προσωπικού πρέπει να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Είναι κατά αποκοπήν στις προτάσεις Κομισιόν. Τώρα, εταιρική σχέση. Συμφωνία σε εταιρική σχέση. Ε, ίσως χρειαζόμαστε πιο σαφή στοιχεία και για να δούμε κυρίως πώς συνδέεται, συνδέονται αυτές τις προτάσεις με τις προτάσεις για τα άλλα ταμεία. Αυτά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ως συμπέρασμα από το εξής για τους δείκτες. Η κατανομή αυτή τη στιγμή βασίζεται, η των βασίζεται στην πυκνότητα, πληθυσμιακή πυκνότητα της κάθε περιφέρειας. Ίσως θα έπρεπε να διαβριθούν λίγο οι δείκτες που έχουμε διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοφέρειας. Για παράδειγμα, γύρανση του πληθυσμού. Ίσως θα πρέπει αυτό το φαινόμενο να συμπεριληφθεί ως ένας δείκτης. Θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις σας τώρα για να βελτιώσουμε την έκθεση και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Είχα πολύ, είχα πολύ καλές επαφές με τους κοιόδης εισηγητές για τη σύνταξη του εγγράφου. Ευχαριστώ. Όσοι μιλήσουν, να μην ξεπεράσουν τα 2,5-3 λεπτά το πολύ. Η Έρικα Μαν έβαλε 7 λεπτά. Σας παρακαλώ να σταθείτε στα πιο σημαντικά για σας, ούτω ώστε να επιτρέψετε και στους υπόλοιπους να πάρουν τον λόγο. Έχω κλείσει τον κατάλογο, έχουμε ένα σκιώδη εισηγητή Μία σκιώδη συγγήτρια. Τον σκιώδη συγγήτρια, τον Φραντσέσκο. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, να, σεβαστώ το χρόνο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά προσπαθώ. Λοιπόν, συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνδεθούμε με το γενικό κανονισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για να αποφύγουμε επικαλύψεις και συγχύσεις αρμοδιοτήτων, και ρόλων. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε για την εδαφική συνεργασία και πρέπει να επιβάλλουμε ένα σύστημα που επιτρέπει ε, την ανταλλαγή πληροφοριών σε πολλά επίπεδα, χωρίς όμως να ξεχάσουμε την απλούστευση, τη σύνθεση που, ζητούμε, που ζητούν οι συνεισηγητές από το Γενικό Κανονισμό. Τώρα μπαίνω στα στοιχεία τα οποία έβαλε η εισηγήτρια. Εκτιμώ τη δουλειά της. Γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένη. Πολύ ακριβής. Συμφωνώ με αυτό το 7%. όχι μόνο ε, για την ευθυγράμμιση με την εκθεση Σάντσε Σμιθ, αλλά το βασικό είναι η πρόταση της Κομισιόν να μην τιμωρήσει την εδαφική συνεργασία, όπως κάνει με άλλους στόχους, φερειπίν τη σύγκληση. Αν θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτό το στόχο και αυτούς, αυτές τις φιλοδοξίες που είχαμε υπόψη μας αρχικά, θα πρέπει να προβλέψουμε μια μεγαλύτερη οικονομική προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των θεματικών προτεραιοτήτων, θα πρέπει η εδαφική συνεργασία να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και να είναι ισότιμη με τους άλλους στόχους. Δεν θα πρέπει δηλαδή η συνεργασία να ξεχνάει τους άλλους στόχους. Θα πρέπει να υπάρχει ε, συνέπεια με το στρατηγικό πλαίσιο, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ε, προκειμένου. Ένα άλλο θέμα αφορά την ευελιξία. Το κριτήριο της ευελιξίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να μπούμε και σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θέλω να καταλάβω πώς η ευελιξία επηρεάζει συνολικά τους στόχους και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Έπειτα, για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Εάν θέλουμε να λειτουργήσουν αυτές, νομίζω ότι η εδαφική συνεργασία δεν μπορεί να είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης. Θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε οι μακροπεριφέρειες να έχουν δικό τους κεφάλαιο. Οι, στρατηγικές, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, ε, είχαν ένα πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη, μια πολλαπλασιαστική επίπτωση. εκφράζουν την ε, μόνιμη συνεργασία μεταξύ λαών ε, και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα και την απλούστευση των διαδικασιών επιλεξιμότητας, συμφωνώ με την εισηγήτρια, θα πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και το γραφειοκρατικό άχθος και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, φορείς που δραστηριοποιούνται σε εδαφικό επίπεδο. Τέλος, για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται και στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας. Ερώτηση είναι αυτή. Γιατί η εδαφική συνεργασία δεν είναι ένας άσχετος στόχος με τους άλλους δύο στόχους του συστήματος της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι μπορούν να ισχύουν και οι ίδιοι κανόνες και εδώ. Αλλά δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Περιμένω τη συζήτηση. Θέλω να θέτω όλα αυτά τα θέματα για να συνεισφέρω κι εγώ στην προσπάθεια της εισηγήτριας. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ε, όλα αυτά τα θέματα. Τέλος, κλείνω και ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για τη δουλειά της. Θα μπω και σε περισσότερες ε, και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες όταν η συζήτηση για το γενικό κανονισμό έχει προχωρήσει, θα έχει προχωρήσει περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λαμπέρ Φανίστερ Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Έχω ένα σημείωμα του Σάντζε Σμιτ ε, και θα τηρήσω τα δυόμιση λεπτά. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σημείωμα. Απαντάει δηλαδή στο έγγραφο εργασία και θέλω από αυτό το σημείωμα να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, για την μακροπεριφερειακή στρατηγική. Καλό είναι να μπουν οι βάσεις αυτής της συνεργασίας ή που έχουν μπει οι βάσεις αυτής της συνεργασίας. Ούτως ή άλλως να προωθηθεί η εδαφική συνοχή. Αυτή είναι η βάση, η εδαφική συνοχή. Χαίρομαι που διάλεξαμε αυτό το σημείο αφετηρίας. Έτσι χρησιμοποιούμε. Αυτό ξεπερνάει όμω του πόρου που έχουμε για του στόχου 3. Πρόκειται για το σκεπτικό γενικά τη περιφερειακή ε, συνεργασία. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. <clears throat> Μετά. Τα τέσσερα αυτά σημεία. Περίεργο που πρέπει να καταλήξουμε σε τέσσερα σημεία. Μήπω θα ήταν να, καλύτερα να ακούσουμε τι αντιδράσει των περιφερειών. Γιατί η διαμεθοριακή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των πολιτών, η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των άνω. Αν υπάρχουν θεματικά ε, κεντρικά σημεία, τι να σας πω. Ίσως χρειάζεται και κάτι συμπληρωματικό που αφορά ακριβώς συγκεκριμένη συνεργασία. Πέρα από τα σύνορα, μεταξύ των υπηρεσιών, μεταξύ των επιχειρήσεων, μεταξύ των σχολείων. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει εκ των κάτω προς τα άνω. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από πάνω. Αυτό με ανησυχεί. Αναφέρθηκε κάτι 7%. Ωραία. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Είναι κίνητρο το 7%. Τι σημαίνει ακριβώς το 7%. Γιατί το είχαμε δεχθεί στην έκθεση πίπα. Εντάξει. Ευχαριστώ Λομπέρ. Γεια Ματούλα. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc ε, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Λάμπερτ, Φανίστερο, είπε ότι το 7% είναι δεδομένο. Αλλά πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό το 7%. Συμφωνώ ότι η ευελιξία πρέπει να αυξηθεί και ότι πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την τοπική αυτονομία, τις τοπικές αρχές, τις τοπικές αποφάσεις αποφάσεις κοντά στους πολίτες και μου φαίνεται ασυνήθιστο να θέτουμε εδώ πέρα γενικούς στόχους τους οποίους επιβάλλουμε εκ των άνω, από αφιψηλού. Να σας δώσω μόνο ένα συγκεκριμένο τομέα ε, ως παράδειγμα για να σας δείξω ότι υπάρχουν διαφορές από τη μία και από την άλλη μεριά των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι πολύ δύσκολο να βάζουμε έτσι αφιψηλού ο, ο, και εκ των άνω όρους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν δρόμοι που περνάνε τα σύνορα, έτσι. Και υπάρχουν από τη μία και από την άλλη μεριά των σύνορων. Δύο χιλιόμετρα, ας πούμε. Τέτοιοι δρόμοι στην Δυτική Ευρώπη Τα δύο χιλιόμετρα μάλλον υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη. 50 χιλιόμετρα είναι το μήκος στην ε, Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πολύ πιο μακρύς, ε, ούτως ώστε να μπορούν οι τοπικές αρχές ανάλογα με τις ε, ανάγκες τους να παίρνουν αποφάσεις. Πρέπει να υπάρχει απλούστευση πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις οι τοπικές αρχές ή θέλουμε να τις επιβάλλουμε τις αποφάσεις αυτές εκ των, άνω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα και αυτά τα project που είναι και τα πιο φθηνά, ίσως είναι και τα πιο πετυχημένα, γιατί επιτρέπουν τις καλές πρακτικές να διαδοθούν. Και θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου για τις ιδέες της και για το έγγραφο εργασίας που μας παρουσίασε. Thank you, ε, Ευχαριστώ, Ιώσιφ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για όλα όσα μας είπε. Ειδικά για τις μακρο περιφερειακές στρατηγικές. Έχω την εντύπωση ότι στο νέο κανονισμό αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και στο μέλλον ε, να βοηθήσουν τόσο ώστε να απτυχθούν οι περιφέρειες. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Πώς θα συντονίσει όλες τις προσπάθειες. Πώς θα ενισχύσει την ανάπτυξη των ε, μακροπεριφερειακών στρατηγικών που κατά τη γνώμη μου είναι εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των περιφερειών και να μπει τέλος στην διαφορά της ανάπτυξης από περιφέρεια σε περιφέρεια. Στο έγγραφο εργασία έχουμε μια αναφορά στο Δούναβι και στη Βαλτική, που είναι περιφέρειες που εντάσσονται σε αυτή τη μακροπεριφερειακή στρατηγική και που είναι πετυχημένα παραδείγματα. Γιατί τα κοινοτικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν και τα, τα κοινοτικά ταμεία χρησιμοποιήθηκαν ε, επιτυχία. Υπάρχει και η περιοχή των Καρπαθίων, πολύ ενδιαφέρουσα επίσης. Ίσως ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και αυτή την ε, περιοχή. Ίσως στην ε, Επιτροπή μας θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τα Καρπάθια που στο μέλλον θα πρέπει να τις δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Σρέντερ. Και εγώ μόνο δύο παρατηρήσεις έχω, μόνο δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Το ένα είναι για τις περιφέρειες της ε, η ε, υπήρχε αυτό το Small Project Fund, ένα ταμείο δηλαδή για μικρά σχέδια. Δεν υπάρχει πια, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το μικρό ταμείο θα πρέπει να διατηρηθεί. Θα ήθελα να ξαναεισαχθεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τομέα γι' αυτό. Μηχανισμοί δηλαδή ιδιαίτεροι για αυτό το ταμείο. Ένα αυτό. Δεύτερον, προς την Κομισιόν. Εντάξει, όλες οι μεθοριακές προ... Ε, περιφέρειες να έχουν την ίδια χρηματοδότηση 75%. Καλή λύση, δεν λέω. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει με εκείνες τις περιφέρειες όπου οι περιφέρειες αυτές αν δεν ήταν στα σύνορα πάνω θα παίρνανε 85% χρηματοδότηση. Ή στην Ελλάδα που υπάρχει μια ειδική κατάσταση 95%. Δηλαδή έχουμε μια περιφερεια που λέει εντάξει εγώ γιατί να ασχοληθώ με αυτό το πρόγραμμα για τα, τις συνοριακές ε, περιφέρειες ε, που θα πάρω μόνο 75% αν κάνω, ακολουθήσω όμως άλλα προγράμματα θα πάρω 85-95% είναι ληστική αντιμετώπιση από τις περιφέρειες ιδίω γιατί δεν έχουν και πολλά χρήματα και δεν θα υπάρχει τελικά μια διαμεθοριακή συνεργασία το πρόβλημα είναι ότι η περιφέρεια αυτή ενδεχομένως δικαιούται για άλλους λόγους υψηλότερα ποσοστά. Και εγώ πιστεύω ότι η διαμεθορική συνεργασία είναι εκείνη που χρειάζεται περισσότερη εργασία και θα πρέπει καν να προβλέψουμε για να ληφθούν υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις που έκανα. Να το ξανασυζητήσουμε δηλαδή πώς θα βρούμε λύση για αυτά γιατί δεν επιτρέπεται άλλες περιφέρειες να έχουν μετά υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης από αυτές που εργάζονται διαμεθοριακά. Ε, τελικά δεν θα γίνει αυτό που θέλουμε. Εγώ δηλαδή ρεαλιστικά όπως τη βλέπω την κατάσταση της περιφέρειας δεν βλέπω πώς θα υπάρχει αυτή η διαμεθορική συνεργασία αν τα ποσοστά είναι τόσο πολύ χαμηλότερα. Ευχαριστώ. Ρίκα, θες να αντιδράσεις? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, πολύ σημαντικές, θα τις λάβω υπόψη. Φυσικά θα γίνει μια έντονη συζήτηση, φαντάζομαι, στο μέλλον, όταν θα μπούμε στο κείμενο και θα το χτενίσουμε. Ήδη μιλήσαμε για κάποια, στοιχεία, για του κειμένου και είδαμε ότι σε πολλές παρεμβάσεις είναι σημαντικό, οι ομιλητέ είπαν ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε τη κάθε περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια θα πρέπει να κρατήσει μια κάποια εξουσία και επομένω θα πρέπει οι αποφάσει να λαμβάνονται υπόψη και σε τοπικό επίπεδο, ούτω ώστε να, λαμβάνονται, να μην ξεχνάμε τι ανάγκε της συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση και την ε, υποστήριξη και τη στήριξη των κρατών, θα υπάρξει συζήτηση θα την παρακολουθήσουμε γιατί υπάρχουν προβλήματα ε, επί των οποίων πρέπει να δούμε τι στάση θα πάρουμε. Κομισιόν. Ε, πολλά τα σχόλια. Ελπίζω ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο κάποια στιγμή να τα πούμε. Να εστιάσω στα πιο σημαντικά όμως. Σε ό,τι αφορά την, ε, το ρόλο του ΕΠΑ. Την πρόταση μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, να συμπεριλάβουμε και τις υποδομές και τις ε, δραστηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είναι σαφές το κανονισμό, μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε. Είναι θέμα διατύπωσης. Συμφωνούμε μαζί σας πάντως. Τώρα, το θέμα της ευελιξίας. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, η Κομισιόν προτείνει ε, αυξημένα ποσά για την εδαφική συνεργασία γιατί πιστεύει πως ε, πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν, έχει, δεν, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της τρέχουσας περίοδου. Τες δείχνουν ήδη ότι πολλά από τα προγράμματα είναι κατακαιρματισμένα, δεν γίνεται επαρκής εστίαση και συγκέντρωση σε στόχους κλπ. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε το μηχανισμό συγκέντρωση, θεματική συγκέντρωση. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Τώρα, για το θέμα του 6% για την τεχνική συνδρομή. Αυτό πρέπει να το δείτε σε συνδυασμό με το ελάχιστο ποσό που προτείνουμε, 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προγράμματα. Το πρόβλημα του ποσοστού της τεχνική συνδρομής είναι πιο σημαντικό στα μικρά προγράμματα και νομίζω ότι βρήκαμε τη λύση του προβλήματος χωρίς να δαπανούμε υπερβολικά ποσά σε δραστηριότητες που ε, δεν είναι αποδοτικές. Τώρα, για το θέμα των εξωτερικών συνόρων. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώ, δεν μπορούμε να το λύσουμε σε αυτόν τον κανονισμό. κοιτάξετε το συνολικό πακέτο, για παράδειγμα τον κανονισμό ENI, και θα δείτε πώς μπορεί να λυθεί αλλού όμως. Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ε, κατανομής, ε, την πληθυσμιακή βάση κλπ. Εξετάσαμε και άλλα κριτήρια, αλλά ε, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία διαθέσιμα για τα διασυνορικά προγράμματα. Το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα. Τώρα, για την συνεισφορά των παραδοσιακών προγραμμάτων, των κλασικών προγραμμάτων. Αυτό ήδη προβλέπεται στον κανονισμό κοινών διατάξεων, ε, ιδιαίτερα μέσω των συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Νομίζω ότι μπορούν να συνεισφέρουν τα παραδοσιακά προγράμματα, ιδιαίτερα μέσω ε, των μακροπεριφερειών και για τα προγράμματα που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες λεκάνες. Στρατηγικές που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες λεκάνες. Τώρα, για τα δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν για το ζήτημα των πρωτοβουλειών μικρών ομάδων διασυνοριακά. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι ανοιχτή σε τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης όπως και στην τρέχουσα περίοδο δυνάμει του άρθρου 6 είναι δυνατόν να προωθηθεί η νομική και διοικητική συνεργασία, αλλά και η συνεργασία ανάμεσα σε πολίτε και φορεί διασυνοριακά. Νομίζω ότι καλύπτονται λοιπόν αυτέ οι δραστηριότητε. Τώρα, για το θέμα του 75%. Είναι περίπλοκο. Η Κομισιόν πρότεινε αυτό το οριζόντιο ποσοστό συγχρηματοδότησης για λόγους απλοποίησης καταρχήν αλλά και διότι ε, δείχνει και τις προθέσεις μας. Η κυρία Στρέντερ μίλησε για τον ανταγωνισμό. Κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Μιλούμε για διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Η, ε, τα προγράμματα επενδύσεων και απασχόλησης ε, έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Για τα διασυνοριακά προγράμματα ε, έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένες διασυνορικές πολιτικές που δίδουν ωφέλη και από τις δύο μεριές των συνόρων. Συνεπώς δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τύπων προγραμμάτων. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε 20 λεπτά για τις υπόλοιπες δύο γνωμοδοτήσεις. Βίκτορ Μποστινάρου. Ταμείο Συνοχής. Περνάμε στη δική του έκθεση. Βίκτορ. τον, ε, στην πρόταση καινούργου κανονισμού θα δείτε αν έχετε διαβάσει το έγγραφο εργασία, ότι πρόκειται για μια σύνοψη των προβλημάτων και των ανησυχιών που εξέφρασαν πολλοί από εσά τις τελευταίες εβδομάδες. Συνεπώ, δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Ε, έχουμε το θέμα των 10 δισεκατομμυρίων που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής στην ε, διευκόλυνση Connecting Europe. Είναι καλή ιδέα, επαναλαμβάνω είναι καλή ιδέα. Δεν διαφωνώ, δεν είμαι αντίθετος με την διαδικασία συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι κάτι που χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνοχή, καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Όμω, οι πολίτες μας και η εσωτερική αγορά χρειάζονται περισσότερο, περισσότερο συντονισμό και καλύτερη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποδομών, ε, είτε είναι ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, είτε είναι μεταφορών. Όπως έχω πει όμω πολλέ φορές, πιστεύω πως χρειαζόμαστε περισσότερες εγγύσει ότι θα γίνουν σεβαστά τα εθνικά όρια προπολογισμών πρόταση λέει πως θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στα, σε project που σέβονται την εθνική κατανομή, την εθνική, του, τους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, που έχουν προβλεφθεί. Αυτό είναι πολύ ασαφές όμως, κατά την άποψή μου. Επίσης δίνει σημαντική υπερβολική ευχέρεια στις ε, φορείς που θα διαχειρίζονται από τις Βρυξέλλες την, ε, το Connecting Europe. Νομίζω ότι αυτό είναι προβληματικό και πολλοί συνάλφοι ε, συμφωνούν. Τα ίδια προβλήματα και τα ίδια ερωτηματικά τα έχουν εκφράσει και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση από την Κομισιόν. Επίσης η Κομισιόν είπε ότι θα εφαρμοστεί η αρχή του First come, first served. Τα πρώτα project που θα υποβληθούν θα είναι τα πρώτα που θα εξυπηρετηθούν. Τώρα μας λένε ότι δεν θα γίνει έτσι, αλλά θα ακολουθηθεί διαφορετική τακτική για αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά δημιουργούν σύγχυση. Η Κομισιόν δεν είναι σαφής ακόμα για το πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις. και πώς θα ε, καθυσυχαστούν οι ανησυχίες μας. Επίσης χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Movement και τη Γενική Διεύθυνση Regio γιατί η διευκόλυνση Connecting Europe έχει σχεδιαστεί από την DG Move, από τη Γενική Διεύθυνση Move, αλλά δεν βλέπουμε τη συνεισφορά της Γενικής Διεύθυνσης Regio. Στο έγγραφο εργασία θα δείτε και κάποιες προτάσεις για το άρθρο 2 που περιλαμβάνει, περιγράφει το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Συνοχή. Ε, ενεργειακή αποδοτικότητα και χρήση ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια σε σπίτια γίνονται επιλέξιμα, ε, επιλέξιμες δράσεις, αλλά ε, αυτό το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή ότι γίνεται επιλέξιμη, γίνονται επιλέξιμες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα σπίτια, ε, θα έχει ε, πολύ σημαντικές συνέπειες. Η ενεργειακή αποδοτικότητα σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αν αυτό συνδυαστεί με αυξημένη χρήση των ενώσιμων πηγών ενέργεια, πραγματικά ευθυγραμμιζόμαστε με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Και μην ξεχνάμε και τα ωφέλη που θα προκύψουν για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και συνεπώ για την κοινωνική διάσταση της οικονομ... και, την... και την οικονομία. Συνεπώ, ε, θα δημιουργηθούν καλύτερε και περισσότερε θέσει εργασία. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο σε πολλέ χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν καλύτερη ε, πρόσβαση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ενέργειας. Αυτές οι επενδύσεις γίνονται... Ε, αν αυτές οι επενδύσεις γίνουν επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, δεν είναι αντιφατικό, δεν δημιουργεί προβλήματα γιατί μέσω του Ταμείου Συνοχής δεν, έχουν, δεν έχουμε χρηματοδοτήσει πολλά τέτοια project. Δεν νομίζουμε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Η άλλη πρόταση που προέκυψε από πολλές συζητήσεις έχει σχέση με την ε, υποστήριξη δράσεων για την μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε δραστηριότητε που περιλαμβάνονται από την οδηγία, καλύπτων την οδηγία 2003 το 87. Το Ταμείο Συνοχής δεν θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί τέτοιες ε, εγκαταστάσεις που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές σε πολλές χώρες του Ταμείου Συνοχής και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα εκπομπές και βέβαια σε επίπεδο του τελικού καταναλωτή. Η υπάρξη χρηματοδότηση αυτών ε, θα είναι πλήγμα για το περιβάλλον και για την Ατζέντα 2020. Σε ό,τι αφορά το 3, ε, είναι πολύ θετική η συμπερίληψη της ενίσχυσης το, της θεσμικής δυνατότητας, θεσμικών ικανοτήτων αναφέρεται, αλλά με γενικά λόγια πρέπει να γίνει πιο σαφής η αναφορά. Ε, θα αναφερθώ στα διδάγματα της ελληνικής εμπειρίας, τα διδάγματα της Ρωμανίας και της Βουλγαρίας και άλλων και θα πρέπει να βελτιώσουμε την, τις διοικητικές ικανότητες, το διοικητικό μηχανισμό όλων των χωρών ακόμα και στο πλαίσιο του Connecting Europe. Πώς σχεδιάζουμε μεγάλα project. Χρειαζόμαστε ε, ικανό προσωπικό, κατηρτισμένο προσωπικό, γιατί υπάρχουν πολλά θεσμικά και διοικητικά προβλήματα. Θα πρέπει ε, τις διοικητικές ικανότητες και τις θεσμικές ικανότητες να τις βελτιώσουμε πριν το 2014, γιατί από το 2014 και μετά θα πρέπει να είναι έτοιμο το προσωπικό που θα χειριστεί αυτά τα προγράμματα να, για να μπορέσουν να αποδώσουν στο 100% των ικανοτήτων τους. Ο Γενικό Διευθυντή κ. Μπέρκοβιτ μου είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει ιδιαίτερη, διάστα... σημασία σε αυτή τη διάσταση. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Για τι άλλε τώρα θα πρέπει ασφαλώ να σεβόμαστε τι ε, διατάξει συνθήκε, αλλά θα πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε ε, βλάβε θα αποφευχθούν. Δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχή θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί όταν ο, ε, ο Ριπένον δεν πληρώσει για την αποζημίωση των ζημιών που έχει προκαλέσει. Είμαι υπέρ τη αρχή ο Ριπένον πληρώνει και είμαι υπέρ υπέρ του το Ταμείο Συνοχής να μπορεί να εμπλακεί σε περίπτωση ε, που ο Ριπένων δεν πληρώσει. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι η οριακή λύση, η τελευταία λύση. Και ο Επίτροπος μου είπε ότι θα λάβει τα μέτρα έτσι ώστε να αποφύγουμε τη, ρήμανση, τη ρήπανση, αν συμβεί ρήπανση ο να πληρώνει και μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσει να εμπλέκεται το Ταμείο Συνοχής για να ε, πληρώσει ε, ρήπανση, οποιαδήποτε ρήπανση ε, μεγάλη διάσταση. Τώρα για την αρσιμότητα. και το Ελεκτικό Συνέδριο ε, χτες και πολλές φορές μας έχουν πει ότι οι κυρώσεις ε, ε, επικαλύπτονται με άλλες διατάξεις και είναι μη αποδεκτές διότι μην ξεχνάτε τα εξής. Έχουμε και την επιστολή των 7 κρατών μελών που και στο Κάγκρε που ζητούν σημαντική μείωση του προπολογισμού του, της πολιτικής συνοχής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα αδειάσει από οποιοδήποτε νόημα είχε. Οπότε θα σε ακούσω και τις γνώμες σας, θα τις ε, λάβω υπόψη μου έτσι ώστε να μιλήσουμε με μία φωνή δυνατόν. Για να εξασφαλίσουμε πολιτική υποστήριξη και στην υιοθέτηση της νομοδότησης στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έτσι ώστε να είμαστε ισχυροί στη διαπραγμάτευσή μας με το Συμβούλιο. Yeah. Ε, ευχαριστώ. Now, uh, Παρακαλώ κύριε Κοτσίσκα, όχι πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ, ε, όλοι οι μελτές. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να πω ότι ελπίζω ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων και ότι δεν θα υπάρχει μείωση του ταμείου αυτού συνοχής. Γιατί ομολογώ ότι όλα αυτά τα ταμεία έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη την ε, ανάκαμψη στα διάφορα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν καλά να το σκεφτούμε το θέμα. Μία μικρή παρατήρηση όσον αφορά το κανονισμό αυτό για το Ταμείο Συνοχής. Ε, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει πλήρη ανάλυση γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν όλα τις ίδιες ανάγκες ή το ίδιο δυναμικό ανάπτυξης. Ας πούμε, οι 12 καινούριε χώρες μέλη έχουν τεράστιες ανάγκες όσον αφορά παραδείγματος χάρη στις υποδομές. Και συμφωνώ με όλους εκείνους που τονίζουν την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος, τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία με λίγες εκπομπές, προστασία του κλίματος, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και ένα άλλο στοιχείο Εκτός από τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ετών, ε, κρατών συγγνώμη, που πρέπει να καλύψουν τα κενά, την καθυστέρηση που έχουν από άλλες χώρες όσον αφορά την οικονομική τους ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν ε, στις χώρες αυτές αυτά τα χρήματα να μπορούν να επενδύονται κατά δυνατόν ευέλικτα. Δεν υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες δηλαδή. Ξέρουμε βέβαια ότι αυτό το ταμείο έχει καταρχήν στόχο την χρηματοδότηση της αηφόρου ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να δώσουμε καταρχήν τη δυνατότητα στις χώρες για να έχουν ανάπτυξη, να κλείσουν το κενό που τους χωρίζει από τις άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι επενδύσεις ε, ε, να έχουν τη δική τους προτεραιότητα μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο, αγαπητέ συνάδελφε Παστινάρο. Η καλύτερη προάσπιση της πολιτικής συνοχής είναι ότι στη σημερινή περίοδο θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που διατίθενται. Αυτό θα πρέπει να είναι το αποδεικτικό στοιχείο. Αλλιώ θα δούμε ότι σε ορισμένες χώρες Ακόμα μάλιστα και στην ηγεσία της Κομισιόν υπάρχει η πρόθεση οι αυτή από την πολιτική, από την ε, πολιτική ε, συνοχής και ανάπτυξης να μεταφερθούν σε άλλους τομείς θα πρέπει να φροντίσουμε και μετά το 2017 να έχουμε ακόμα χρήματα για το Ταμείο Συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να ασχοληθείτε με κάθε συνέπεια στην εφαρμογή και επίτευξη αυτών των στόχων. Δεύτερον, και αυτό αφορά επίσης από τη θεματική χρήση της ενέργειας και ε, την ε, κατασκευή κατοικιών. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η απορρόφηση είναι πάρα πολύ μικρή Δηλαδή αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει οι στόχοι που έχουν ήδη καθοριστεί, τα χρήματα που έχουν ήδη προβλεφθεί να χρησιμοποιούνται. Connecting Europe, συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν, αλλά έχω ακόμα περισσότερες. Γιατί δεν θέλουμε εδώ να έχουμε απλώς μια αρχή χρηματοδότησης, αλλά η αρχή αυτή θα πρέπει να έχει επίδραση και στον προγραμματισμό εκεί που σε ορισμένα κράτη-μέλη, στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα ε, σύστημα προγραμματισμού που αρχίζει από το ομοσπονδιακό επίπεδο και φτάνει μέχρι το τοπικό. Λοιπόν, θα πρέπει πριν έχουμε μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις να γίνει η συζήτηση για την ε, πραγματοποίηση των στόχων όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές και μάλιστα στον τομέα παραδείγματος χάνης της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας που έχει ένα ρόλο να παίξει. Και αυτή η αρχή για την σύνδεση δεν θα μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να παίξει το ρόλο της, οπότε τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση θα κάνω μόνο. Θέλουμε να επιμείνουμε στο εξής. Θα πρέπει στο μέλλον να επενδύσουμε πολύ στις υποδομές και κυρίως στις ερευνητικές υποδομές. Δεν μιλάω για, την, για τον πετόν και την άσφαλτο, έτσι, αλλά μιλάω για τις εγκαταστάσεις, για τις υποδομές. Η Επιτροπή Ήτρε, στα πλαίσια του Horizon, είπαμε ότι πρέπει ή μάλλον ότι είναι απαράδεκτο το 80-90% των διαθέσιμων πόρων να πηγαίνουν συνέχεια στα ίδια κράτη-μέλη επειδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι απαράδεκτο. Τι πρέπει να κάνουμε κύριε Μποστινάρου, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Περιβάλλον, ναι φυσικά, αλλά και υποδομές, ερευνητικές υποδομές. Θα πρέπει να επενδύσουμε μαζικά σε αυτές τις υποδομές. Και σε επίπεδο κρατών μελών αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να έχουμε ευκαιρίες ούτω ώστε να υπάρχει μια επανεξισορρόπηση της κατάστασης στην Ευρώπη. Ε, αυτός είναι ο στόχος. Όταν μιλάμε για εδαφική συνοχή πρέπει να επενδύουμε μαζικά σε αυτό το στόχο της συνοχής. Αλλιώς θα κάνουμε ένα ιστορικό λάθος. Πρόεδρος. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Μποστινάρου, και μετά η Κομισιόν, γιατί θέλουμε τελείωσαν οι ομιλητέ. Ναι, να απαντήσω πολύ σύντομα σε κάποιε από τις παρατηρήσεις. Φυσικά συμφωνώ ότι τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά και το ποσοστό απορρόφησης θα πρέπει να αυξηθεί δραματικά. Φερρυπίν η χώρα μου είναι ο χειρότερος μαθητής στην Ευρώπη και η επόμενη, αμέσως επόμενη είναι η Βουλγαρία. Αλλά εγώ δεν μιλάω για την δική μου περίπτωση, τη Ρουμανία. Αλλά εγώ μιλάω για τη φιλοσοφία, για, τη, για τις αρχές που πρέπει να διέπουν το σημείο αυτό. Ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόσουν προγράμματα εν ευθέτω χρόνο, ούτως ώστε να μην χάνουν χρήματα. Άρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αύξηση του διοικητικού δυναμικού, ούτως ώστε να αυξηθεί και το ποσοστό ε, απορρόφησης. Κύριε Γιωακίν Τέλερ, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Επίσης η μείωση του χάσματος της ανάπτυξης. Φυσικά αυτή είναι η ουσία της πολιτικής συνοχής. Αλλά με την κρίση, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αυτό το χάσμα αυξάνεται, βαθαίνει ανάμεσα στην ανάπτυξη κάποιων κρατών μελών και κάποιων άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ε, θα πρέπει να υλοποιήσουμε την αρχή. Και έπειτα, εγώ δεν είμαι υπέρ των δεσμευτικών κανόνων. Όχι, εμένα μου αρέσουν οι ευέλικτοι τρόποι πρόσβασης ε, στα κονδύλια και για την ενέργεια. Το ίδιο χρειαζόμαστε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιοχές, τις περιφέρειες. Δεν θέλουμε να βοηθάμε μόνο τους δημόσιους φορείς. Άδειοι εκπρόσωποι των περιφερειών εκφράζουν τις ανάγκες τους όλοι οι συνάδελφοι από την Ανατολική και ε, Κεντρική Ευρώπη είπαν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, τότε πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά που είπαν. Αυτό το μέσο για την ε, σύνδεση της Ευρώπης. Ε, συμφωνώ μαζί σας. Είμαι υπέρ επί της αρχής, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες και τόσα ερωτηματικά στις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέσο σύνδεσης της Ευρώπης, γι αυτό πρέπει να, που γι' αυτό πρέπει να εγγύψουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είμαι σε επαφή με τον κύριο Πίπερ, που είναι ο εισηγητής για αυτό το μέσο, συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, αυτά τα ερωτηματικά δεν τα θέτουν μόνο οι ευρωβουλευτές, τα θέτουν και τα κράτη-μέλη. Ε, χρειαζόμαστε καλύτερες απαντήσεις για να δούμε αν θα δεχτούμε ή όχι αυτό το μέσο, το, Connect, το Connecting Europe για τα κέντρα αριστείας ε, στην έρευνα και στην ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με την ιδέα του κ. Ρόη. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που τα δημόσια κονδύλια στα κράτη-μέλη μειώνται δραματικά. Και ξέρετε τι για ποιο λόγο γίνονται αυτές τις περικοπές. Λόγω της μαγικής λέξης λιτότητα ε, η λιτότητα μπορεί να καταστρέψει την ουσία και το πνεύμα της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ματσόνη μόλις ήρθε. Σας παρακαλώ, άντε, σας δώσω το λόγο, αλλά πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου, που παρεμβαίνω μετά από αυτόν, μετά τη δεύτερη του παρέμβαση. Ένα στοιχείο θέλω να προσθέσω Ίσως αυτό που θα πω το είπε στην πρώτη του παρέμβαση που δεν την άκουσα. Τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την κάλυψη του Ταμείου Συνοχής και σε άλλες περιοχές, πέρα από αυτές που προβλέπονται σήμερα, που είναι οι παραδοσιακές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα καινοτόμου από πλευράς Κομισιόν. Αυτές προβλεπόταν και προβλέπονται. Η θέση που έχω εκφράσει πολλές φορές είναι αυτό το ταμείο να είναι πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό. Και αυτός ο στόχος της μεγαλύτερης παραγωγικότητας για τα κράτη που είναι δικαιούχοι δεν πρέπει να γίνει μέσω επέκτασης των περιοχών και των τομέων όπου παρεμβαίνει το Ταμείο, αλλά χάρη στη μεγαλύτερη ευελιξία των προγραμμάτων που επωφελούνται από πολλά ταμεία. Δηλαδή να είναι πιο συμβατά μεταξύ τους τα διάφορα ταμεία, ούτως ώστε να παρεμβαίνουν και σε διαφορετικούς τομείς, πέρα από τις υποδομές και το περιβάλλον, που είναι οι τομείς που υποφελούνται από το Ταμείο Συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και στο σχέδιο του κειμένου του κυρίου Μποστινάρου κάπου θα πρέπει να μπει και αυτό το σημείο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα σημεία που προβλέπουμε για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το θέμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας των οικοκυριών. Υπάρχουν δύο θέματα. Ε, υπάρχει ένα θέμα αρχής και υπάρχει και ένα θέμα εφαρμογής. Το θέμα της αρχής, καταρχήν. Από πλευράς Κομισιόν θεωρούμε ότι το Ταμείο Συνοχής είναι ο μηχανισμός που έχουμε για τη βασική υποδομή, για τις βασικές υποδομές. Και για να πετύχουμε κάποια πράγματα στο περιβάλλον και στις μεταφορές. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν σημαντικές ανάγκες στα νέα κράτη-μέλη στους τομείς αυτούς. Τώρα, για την ενεργειακή αποδοτικότητα των νοικοκυριών. Όπως είπε ο κύριος Μποστινάρου, είναι επιλέξιμα για υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στην τρέχουσα περίοδο, το, τα ποσά στις χώρες συνοχής είναι ανάμεσα σε, στο 1 και στο 2% του συνολικού ποσού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν νομίζουμε ότι υπάρχει αδύρυτη ανάγκη για να ανοίξουμε το Ταμείο Συνοχής. Γιατί ούτω ή άλλω οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχουν απορροφηθεί πλήρω. Αν φτάναμε στο 5 ή 10% εντάξει θα ήταν ένα επιχείρημα αυτό. Στον τομέα τώρα της ανταλλαγής στο μηχανισμό ETS, ε ανταλλαγής ε, δικαιωμάτων εμπορίας. Έχουμε τον αποκλεισμό ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζονται να επηρεάζει το τομέα CTS ε, ε, της ενέργειας. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την τιμή του άνθρακα. Mm. Δεν θέλουμε να υποσκάψουμε το μηχανισμό εμπορίας εκπομπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην θέρμαση και στη συμπαραγωγή. Υπάρχει ένα θέμα μεγέθους της εγκατάστασης και είδους εγκατάστασης. Αυτές οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά μπορούν να αποφεληθούν. Είναι ένα σημαντικό θέμα για την Κομισιόν. Και μπορούμε να δώσουμε και περαιτέρω τεχνικές ε, εξηγήσεις. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Για τα υπόλοιπα θέματα, χαιρόμαστε για τα σχόλια του εισηγητή για την, το θεσμικό δυναμικό, για την αρχή ο Ριπένον πληρώνει και ελπίζουμε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τη δουλειά που κάνει αυτή η Επιτροπή. Πάμε στο τελευταίο σημείο. Του Γιώχημ Ξέλε για το κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ομιλίο Ευρωπαϊκής Συνεργασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει πολύ προχωρήσει η ώρα και γι' αυτό θα ήθελα να ακολουθήσω τις ε, προτραπές σας να είμαι πολύ σύντομος ε, και ιδίω ως εισηγητής να μην μακρηγορήσω για να μπορούν οι συνάδελφοι να παρουσιάσουν αποφάσει του. Ιδίω μια που στην τελευταία μα συνεδρίαση συζητήσαμε το θέμα του περιεχομένου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Συνεργασίας. Συνεργασία. 18 τέτοιοι όλυμοι έχουν ήδη δημιουργηθεί, έχουν ιδρυθεί. Οι αντιδράσεις αυτών που έχουν ιδρυθεί είναι ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το διευρυμένο νομικό πλαίσιο που παρουσίασε η Κομισιόν τώρα και ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μέσο αυτό για διαμεθορική συνεργασία όπως φαίνεται ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα έχω νέες ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους που θέλουν να θέσουν σε αυτό το νομικό πλαίσιο την διαμεθορική συνεργασία. Νομίζω ότι η συζήτηση σχετική θα μας ακολουθήσει αρκετό καιρό, ιδίως μια που η συνεδρίασή μας τον Απρίλιο προβλέπει μία κρόση των εμπειρογνωμάνων για το θέμα αυτό. Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι ο οικονομισμός για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία δεν προβλέπει συνεργασία με τρίτες χώρες. Έχω να πω ότι αυτό είναι δυνατόν μέσω αυτών των ομίλων που επιτρέπουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και επίσης συνδυασμό με μέσα της ε, πολιτικής γυτνίασης και με στοιχεία της ε, ε, πολιτικής συνοχής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό το νομικό μέσο να γίνει καλύτερα γνωστό και εδώ στο Κοινοβούλιο, στους αρμοδίους συναδέλφους, στις άλλες επιτραπές, γιατί τώρα πια όλες οι πολιτικές και όλοι οι τομείς δράσης των ε, διαχωριστικών πολιτικών μπορούν να καλυφθούν από τα ΕΕΣ. Πολιτική για το ίδρυμα για την ενέργεια κλπ. Οι κύριε συζητήσει θα γίνουν νομίζω με την εφαρμογή των διατάξεων γιατί ορισμένα κράτη-μέλη και ορισμένες περιφέρειες που έχουν πιο ευρία συμφέροντα φαίνεται ότι είναι επιφυλακτικές ε, και επιφυλακτικά τα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτή τη δυνατότητα των μεθοριακών περιοχών να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο. Θα ακούσω με ενδιαφέρον την συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, εγώ ευχαριστώ Γιώργη. Η κυρία Σμόλκοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ξεκάθαρα ότι η Κομισιόν μας έδωσε πολύ καλά ε, έγγραφα για το θέμα αυτό και επίσης θέλω να επενέσω την εργασία του κ. Τσέλερ γιατί το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ ευανάγνωστο και ο στόχος βέβαια είναι η απλούστευση. Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πριν εγγραφεί αυτό το έγγραφο είχαμε μια ευρεία διαφορετική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και όλα τα σχόλιά τους έχουν ε, ενταχθεί σε αυτό το έγγραφο. Οι πιο σημαντικές καινοτομίες της πρότασης έχουν ε, παρουσιαστεί ξεκάθαρα. Αυτό νομίζω είναι προς όφελος όλων, γιατί οι καινοτομίες αυτές στο μέλλον θα διευκολύνουν τη δημιουργία αυτών των ομίλων τοπικής συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε επίσης την κλίση αυτή προς όλες τις χώρες μέλη να ευθυγραμμίσουν τα νομοθετικά τους κείμενα και τις πρακτικές τους με αυτό το σημείο. Γιατί εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε επίπεδο κρατών μελών δηλαδή. Εδώ έχουμε λοιπόν μια δυνατότητα Βελτίωση του εγγράφου. Να συμπρέξουν δηλαδή και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Χρυσμένοβα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όλα όσα ανέφεραν οι συναδελφοί μέχρι στιγμή. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ορισμένα σημεία. Πρώτον, συγχαρητήρια προ την Επιτροπή για τις προτινόμενες ε, τροποποιήσεις του κανονισμού. Βλέπουμε ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα κύρια προβλήματα. Επίσης βλέπουμε τις προσπάσεις που γίνονται για ολοκλήρωση. Η συμμετοχή σε, αυτές, ε, σε αυτούς τους ομίλους συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά παραδείγματος χάρη μη κυβερνητικές οργανώσεις, όσον αφορά τρίτες χώρες, νέα μέλη στους ομίλους αυτούς ενδιαφέρον, το υποστηρίζω, υποστηρίζω την αρχή αυτή και θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα εγγυηθεί καλύτερη ασφάλεια και δυνατότητα προγραμματισμού για τις, τους νέους αυτούς ομίλους συνεργασίας. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να συζητήσουμε το κατά πόσο ήταν καλή ιδέα το να αυξηθεί η εν λόγω χρονική περίοδος τόσο πολύ. Επίσης δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τις ε, ε, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, τους κανόνες δράσης και το συντονισμό. Κατά τα άλλα όμως νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα πρόοδου. Συμφωνώ με τον συγητή τον κύριο Τσέλερ όσον αφορά την ιδέα της ε, μοναδικής θηρίδας ε, για την ε, προσέγγιση. Επίσης χαιρετώ την πρόταση της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογή των ομίλων αυτών γιατί αυτό εντάσσεται στην στρατηγική του 2020. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι οι ευρωπαϊκοί αυτοί ομιλοί για την αρφική συνεργασία έχουν μεγάλο δυναμικό και θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε προσπαθώντας να διατηρήσουμε την ιδέα τους, την ουσία τους και να μην περιπλέξουμε τους κανόνες. Ματούλα. Ιωσήφ Ματούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το συνάδελφο, τον κύριο Τσέλερ, για το έγγραφο που μας υπέβαλε. Είναι ένα πολύ ρεαλιστικό έγγραφο. Μιλάει για πολύ απλά πράγματα που πρέπει να γίνουν με σκοπό την απλού, απλούστευση αυτής της μορφής της οργάνωσης που υπάρχει από το 2007. Αυτές τις εδαφικές ομάδες συνεργασίας. Φυσικά μόλις τώρα έχουν αρχίσει να δουλεύουν ε, και τα μέτρα απλούστευσης είναι ευπρόσδεκτα, γιατί στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση δυσκολεύεται από, την, από το νομικό πλαίσιο και από, τις, ε, τη διοικητική δομή που υπάρχει στα ανατολικά κράτη, που είναι τελείως διαφορετική από αυτό που από την πραγματικότητα που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη. Μπορεί να υπάρχουν τεράστιε διαφορέ ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε μια τέτοια ομάδα, σε ένα τέτοιο όμιλο εδάφική συνεργασία. Την περασμένη Παρασκευή κάναμε μια πρώτη συνάντηση ξεκινήσαμε μία τέτοια ομάδα μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Είχαμε εκπρόσωπους από τα Υπουργεία, από τις περιφέρειες, από, τα, δήμους και τις κοινότητες και φυσικά από την εθνική διοίκηση είπα. Και εκεί ε, ακούστηκαν διάφορα πράγματα που συζητάμε και εδώ σήμερα. Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν αυτές τις διαφορές στην νομοθεσία μεταξύ των ε, συμμετεχόντων. Αν θέλουμε δύο ας πούμε, νοσοκομεία να συνεργαστούν, δηλαδή συνεργασία σε επίπεδο υγείας, έχουμε από τη μία ένα νοσοκομείο ας πούμε, το οποίο το διαχειρίζεται μια τοπική αυτοδιοίκηση και από την άλλη έχουμε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, το οποίο το διαχειρίζεται ε, το κράτος, ας πούμε, ή το, το Υπουργείο δηλαδή. Ε, το πλαίσιο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. Πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε όλα τα προγράμματα και όλα τα σχέδια σε μια διασυνοριακή περιοχή. Α πούμε, ο δρόμο γύρω από το νοσοκομείο, στη μία και στην άλλη περίπτωση, τη μία, στη μία περίπτωση το διαχειρίζεται το κράτο και στην άλλη ε, η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δούμε ποιε είναι προτεραιότητε στο διασυνοριακό επίπεδο. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Φυσικά, όλα τα project δεν, χρησιμο χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορεί, ας πούμε, το, τοπικοί φορείς ή άλλες πηγές να χρηματοδοτούν κάποια project. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να θέσουμε προτεραιότητες, δηλαδή για διασυνοριακά προγράμματα ή διαπεριφερειακά προγράμματα. Ε, θέλω να καλωσορίσω τις νέες ιδέες, ε, δηλαδή τα κριτήρια απόρριψης για πολλαπλές αιτήσει. Ε, πολλαπλή υποβολή του ίδιου προγράμματος ή το One Stop Shop, τη μοναπευθυντική θηρίδα. Στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν τεράστιες διαφορές ό,τι αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να πληρώνουμε τους συμμετέχοντες σε τέτοια project. Ε, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις απολαβές, στους μισθούς. Όταν έχουμε ένα ενιαίο κριτήριο για τη χρηματοδότηση, Μπορούμε και σε προγράμματα διαπεριφερειακά ή διασυνοριακά να έχουμε τέτοια απλά ενιαία κριτήρια που να αφορούν τις χώρες που συμμετέχουν στο project αυτό. Αυτά και ευχαριστώ ακόμα μια φορά τον συνάδελφο τον κύριο Ζέλλερ. Γιωακίμ, θες να αντιδράσεις? Ε, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεισφορά σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που με τονώνετε, έτσι με ενισχύετε. Χάρη στη συνεργασία όλων των συναδέλφων έχουμε ένα καλό έγγραφο εργασία, το οποίο βέβαια πρέπει να το βελτιώσουμε περαιτέρω, για αυτά που είπε ο συνάδελφος Ματούλα, για τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Φυσικά, καταρχάς, ε, χρειάζεται καλή θέληση από όλου από όλα τα επίπεδα και τα κέντρα εξουσίας, όποια και αν είναι αυτά τα οποία συμμετέχουν. Ε, τα αποτελέσματα αυτά τα έχουμε σε τοπικό επίπεδο. υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν ε, ευκαιρίες ε, σε όλα τα επίπεδα, αλλά τα αποτελέσματα είναι σε τοπικό επίπεδο. Ε, Μποστινάρου, η συμβατότητα των κανόνων είναι πολύ σημαντική όταν ε, υπάρχουν τόσα πολλά ταμεία. Η Κομισιόν μας μια διευκρίνηση ότι το Κοινωνικό Ταμείο, το ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κτλ. Θα, όλα αυτά τα ταμεία θα τα διαχειριστούμε με συμβατό και συνεκτικό τρόπο. Οι κάνονες θα είναι οι ίδιοι. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πολυταμιακή. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι αλλοσυγκρουόμενοι οι κανόνες, ε, πρέπει να έχουμε ένα κανόνα σαφή που να έρχεται να ξεκαθαρίζει τι ισχύει. Έπειτα, ένα δρόμο για τι κοινότητε και τις περιφέρειες ε, που εμπλέκονται σε τέτοια προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε το ρόλο των περιφερειών και των τοπικών αρχών ε, στα προγράμματα αυτά, η Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, τον David Sweet. Ευχαριστώ τον Ιωάκιμ για την ε, έκθεσή του αυτή που είναι πολύ άρτια και ε, χρήσιμη. Νομίζω πως όλοι κατανοούμε πως προτείνουμε κάτι που δεν αποτελεί τμήμα του πακέτου συνοχής, ε, τουλάχιστον όχι επίσημα και τυπικά. Δεν κατανέμουμε κονδύλια συγκεκριμένους στόχους είναι ε, μια πρόταση για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και να ελοπίσουμε προγράμματα, διασυνορικά προγράμματα συνοχής. Θα ήθελα να συγχαρώ το κοινοβούλιο που έχει οργανώσει αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι παρόμοιο στο Συμβούλιο. Ελπίζουμε θα το πετύχουμε. Γιατί μέχρι τώρα έχουν συζητήσει πιο σοβαρά μόνο πράγματα συμβουλια. Ε, δεν έχουμε πρόβλημα με τις προτάσεις σας, με τα σχόλιά σας. Για μας πρόκειται για ένα εργαλείο. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας είναι ένα εργαλείο το οποίο όμως μπορεί να χρηματοδοτηθεί ε, χωριστά ε, αφορά μάλλον δραστηριότητε, οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ε, ξεχωριστά αλλά τις φέρνουμε κάτω από την ίδια στέγη. Οπότε θέλουμε να διευκολύνουμε τη χρήση αυτών των, αυτού του εργαλείου χωρίς όμως να το τεντώσουμε υπερβολικά πολύ για να καλύψει δραστηριότητε που, θα που θα, μάλλον θα έπρεπε να καλυφθούν διαφορετικά. Ε, πρόκειται για ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Χαίρομαι που συμφωνείτε με την ιδέα της σιωπηρής έγκρισης γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα για τη δημιουργία τέτοιων ομήλων μέχρι τώρα ήταν οι ε, μακρόχρονες ε, και πολλές φορές αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα αιτήματα δημιουργίας ομίλων. Προφανώς οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν την τελική αρμοδιότητα σύμφωνα με την εθνική Νομοσία και το Εθνικό Σύνταγμα της κάθε χώρας ε, για να εγκρίνουν ή όχι τέτοιες δραστηριότητε. Όμως έχουν και την ευθύνη αν έχουν αντιρρήσεις να τις εκφράσουν έγκαιρα και γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο επιμαχό σημείο του πακέτου. Τέλος, ευχαριστώ πολύ που υποστηρίζετε την διεύρυνση των ομίλων έτσι ώστε να περιλάβουν και τρίτες χώρες. Είναι η αλλαγή που πιο πολύ μας ζητήθηκε από υπάρχοντες ε, και ενδυνάμει μελλοντικούς ομίλους. Ελπίζω ότι θα πιστεί και το Συμβούλιο. Υπάρχουν σίγουρα και τεχνικά θέματα τα οποία θα προκύψουν, και ελπίζω ότι θα επιληθούν. Θα συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες για να συμπεριλάβουμε τις καλύτερες ιδέες μέσα στον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ και για την μέχρι τώρα συνεισφορά σας. Ευχαριστώ, David, λέει πρόεδρος. Ε, τελειώνουμε με την ημερησία διάταξη. Ε, εδώ πέρα θα συναντηθεί η ομάδα εργασίας για την απλοποίηση με τον Νίκολας Μάρτιν κλπ. Είναι μεγάλη αίθουσα, ε, μπορείτε να παρευρεθείτε όλοι. Δεν θα έχουμε βέβαια γεύμα, δεν θα σερβιριστεί, οπότε το έχετε το υπόψη σας. Η επόμενη συνεδρίαση το Μάρτιο 19 και 20 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ.